colleagues, ladies and gentlemen, Αγαπητοί συνάδελφοι, σας καλωσορίζω ε, μετά το μεσημεριανό διάλειμμα ε, να καλωσορίσω μια ομάδα από τη Βουργουνδία ε, οι οποίοι συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα Erasmus Plus και εκπροσωπούν δασκάλους, διευθυντές σχολείων, επιθεωρητές. Σας καλωσορίζουμε θερμά στην Επιτροπή μας. Σήμερα το απόγευμα θα έχουμε μία ακρόση σχετικά με τις πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης, ε, οι προοπτικές που υπάρχουν από αυτού. Έχουμε καλέσει οκτώ εμπειρογνώμονες που σημαίνει ότι θα πρέπει να τηρήσουμε ακριβώς το χρόνο που έχουμε προβλέψει, γιατί θέλουμε όχι μόνο να ακούσουμε τους εμπειρογνώμονες, αλλά να έχουμε μετά και χρόνο για ερωτήσεις και να δοθούν και απαντήσεις. Παρακαλώ λοιπόν, όχι μόνο οι εμπειρογνώμονες ε, να τηρήσουν το χρόνο, αλλά και οι συνάδελφοι να μην βγάζουν λόγους, αλλά να κάνουν συγκεκριμένες ερωτήσεις, γιατί σήμερα αυτό που ενδιαφέρει είναι να ακούσουμε τους εμπειρογνώμονες και ελπίζω μετά να έχουμε μια ιδιαίτερα ζωντανή συζήτηση. Από το 1985 κάθε χρόνο έχουμε τουλάχιστον δύο πρωτεύουσες στην Ευρώπη, οι οποίες επιβραβεύονται ως ε, πρωτεύουσε της Ευρώπης και ο στόχος σε αυτή την περίπτωση είναι να ανανεωθεί η πόλη, να αλλάξει η εικόνα της πόλης ε, και να ε, προβάλλονται πολιτιστικές εκδηλώσεις και προς τα Ο στόχος είναι ο πολιτισμός με την ευρύτερη έννοια, γιατί αυτό που ενδιαφέρει είναι να υπάρξει και μια βιώσιμη εξέλιξη της πόλης. Άρα δηλαδή όχι μόνο να έχουμε κάποιες εκδηλώσεις και κάποια φεστιβάλ μιας μέρας. Όχι, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Μας ενδιαφέρει να δημιουργήσουμε δίκτυα που θα βελτιώσουν τον πολιτισμό στις πρωτεύουσες. Κατά τη διάρκεια όλων των ετών, οι πολιτιστικέ πρωτεύουσες τη Ευρώπη υπογράμμισαν τον πλούτο της Ευρώπη που επιτρέπει στους Ευρωπαίους πολίτες να αποκτήσουν την αίσθηση του ότι ανήκουν σε ένα κοινό πολιτισμό και μπορούν να εορτάζουν τα τοπικά τους ήθη και έθιμα. Οι ε, πόλεις πολύ συχνά εκμεταλλεύονται αυτή την ευκαιρία για να νεωθούν, για να αναπτύξουν το δυναμικό τους και για να αναπτύξουν νέε φόρμες νέες μορφές του τουρισμού. Ε, το να είναι μια ε, πρωτεύουσα, πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης μπορεί να βοηθήσει την κοινωνική συνοχή και μπορεί επίση να προβάλλει και τον ρόλο των πολιτών στην πόλη, τους δίνει και τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε πολιτιστικές εκδηλώσεις. Τα θέματα που έχουν σχέση με τις πολιτιστικές πρωτεύουσε και ενδιαφέρουν εμά ως ευρωβουλευτές, θέματα τα οποία μπορούν να απαντηθούν σήμερα από τους εμπειρογνώμονες, είναι ερωτήματα όπως παραδείγματος χάρη, ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των προγραμμάτων, ποια ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία, ποιε ήταν οι ε, προεκτάσεις διαρκείας. Το θέμα της κληρονομιάς είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και στις δικές μας συζητήσεις. Ε, πώς πρέπει να είναι η πολιτιστική πρωτεύουσα, πώς άλλαξε μία πόλη. Οι εμπειρογνώμονες, ε, αν μας πούν κάτι άλλο, θα ήταν λάθος. Είπαμε ότι ε, πρέπει να μιλήσουμε και για λάθη. Ε, με τον τρόπο αυτό μπορούμε να αποφύγουμε τα λάθη και ως εκ τούτου μπορούμε να μάθουμε όχι μόνο από τα δικά μας αλλά και από τα λάθη των άλλων. Ε, το ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσον υπάρχει μια στρατηγική για τον βιώσιμο τουρισμό και ποια συμβουλή θα δίνατε στο μέλλον στα δημοτικά συμβούλια. Οι πολίτες εντάσσονται σε αυτή την πρωτοβουλία ή υπήρξαν περισσότερο θεατές. Άλλο ερώτημα, ποια ήταν η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Η ε, πόλη σας συνεχίζει να συνεργάζεται με τις υπόλοιπε πολιτιστικές πρωτεύουσες. Υπάρχει ένα δίκτυο, ε, το πρόγραμμα των ευρωπαϊκών πολιτιστικών πρωτεύουσων, μήπως πρέπει να ανανεωθεί και να προσαρμοστεί. Αυτό θα πρέπει πρέπει κατ' ουσία να είναι το οδηγό νήμα εκείνων που θα ακούσουμε σήμερα. Η ακρόση αποτελείται από δύο τμήματα. Στο πρώτο κομμάτι ε, θα ακούσουμε τους διευθυντές, τους μάνατζερ που θα μιλήσουν για την εμπειρία τους και κατά το δεύτερο κομμάτι της εκδήλωσης ε, θα έχουμε τα μέλη ε, του Συμβουλίου Αξιολόγησης που θα μας παρουσιάσουν και εκείνη την εμπειρία τους. Έχουμε καλέσει καταρχήν τον κύριο Χαβιέ Φιντέλ Παρουής, ε, πρώην καλλιτεχνικό διευθυντή του Ιδρύματος ε, για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα στο Σαν Σεμπαστιάν το 2016. Μετά, ε, Ζήρι Σουτσάνεκ, πρώην διευθυντής του Πίλσεν, Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα, το 2015, όπου πήγαμε κιόλα με την Επιτροπή μας, κατόπιν Τάμα Σαλάι, πρώην Διευθυντής της Πολιτικής Ένωσης του ΠΕΣ το 2010 και η κυρία Διάννα Σίπτσεπε, ε, πρώην ε, καλλιτεχνική διευθύντρια ε, του προγράμματος στη Ρίγα το 2014 και τέλος, εξίσου όμως σημαντική, η κυρία Ροσέλα Ταραντίνο. Όσοι ήταν μαζί μας σήμερα στη Μαδέιρα ε, θα την γνώρισαν ε, και θα διαπίστωσαν το πόσο ενθουσιασμένη είναι για την πολιτιστική πρωτεύουσα Μαδέιρα. Έχουμε και την κυρία Σίμια Άμαν και Βλάζεκ ε, που είναι μέλη του Συμβουλίου Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας και την κυρία Μπεατρίς Γκαρσία, την οποία ε, Όρη η Επιτροπή και με την οποία έχουμε ήδη συνεργαστεί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα όλοι εδώ, ε, που είστε στη διάθεσή μας για ερωταπαντήσεις. Για μας αυτό που έχει σημασία είναι να μπορούμε να ανταλλάξουμε απόψεις, έτσι ώστε να διαμορφώσουμε τις μελλοντικέ μας εργασίες και σε τελική ανάλυση τις εμπειρίες σας να μπορέσουμε να τις συμπεριλάβουμε στη δουλειά μας. Θα ήθελα για άλλη μια φορά να επισημάνω ότι έχουμε χρόνο ε, αγόρευσης περίπου 7 λεπτών για κάθε εμπειρογνώμονα και θα ήθελα να δώσω ε, πρώτα απ' όλους το λόγο στον κύριο Χαβιέ Φιντέλ Πάγια Ρουής. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Είναι έτοιμη η παρουσίασή μου, ρωτάμε ο μιλητής. Αξιότιμα μέλη της Επιτροπής αυτής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε σε αυτήν τη συνάντηση. Για μένα είναι μεγάλη ευθύνη και μεγάλη τιμή που επιλέχθηκα ανάμεσα στους διάφορους καλλιτεχνικές ε, διευθυντές, οι οποίοι έχουν δουλέψει από το 1995. Είναι μεγάλη η ευθύνη για μας να κατανοήσουμε ότι πρέπει να είμαστε σε θέση να προσαρμόσουμε το πρόγραμμα. Είναι ένας ε, αγώνας βέβαια ε, να λάβουμε υπόψη μας όλες τις διατερότητες της ευρωπαϊκής ε, ε, κουλτούρας μέσα σε 7 λεπτά. Προσπάθησα να φτιάξω μια αλφάβητο με γράμματα που μπορεί κανείς να καρφώσει. Και βάσει αυτών έχω φτιάξει 26 ιδέες κλειδί. Πρώτον, από το α, agreement, συμφωνία. Θα έπρεπε μια πόλη να είναι υποψήφια αν δεν έχει τη στήριξη σε εθνικό επίπεδο ή τουλάχιστον που να δέχεται το κοινό την υποψιότητα αυτή. Αλλιώς μήπως δεν θα έπρεπε να δοθεί υποψιότητα αυτή αν κάποια πόλη θεωρεί ότι τιμωρείται με το να γίνεται πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Αυτό θα πρέπει να το αποφύγουμε βέβαια. B. Behavioral change. Θα πρέπει οι πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης να δημιουργούν κάποια αλλαγή στην ζωή των πολιτών, να να καταλάβουν καλύτερα την Ευρώπη για παράδειγμα. Έπειτα, C. Culture. Ποια όμως ε, culture, για ποια κουλτούρα μιλάμε, πώς αυτή καθορίζεται και πώς την κατανοούμε. Ε, τι, σε τι αξίες ε, βασίζεται τις κοινέ των Ευρωπαίων βέβαια που μας κάνουν να αισθανόμαστε όταν ανήκουμε στον ίδιο κοινό χώρο. Νομίζω ότι οι πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης θα πρέπει να αποτελεί το εργαλείο που επιτρέπει στον κόσμο να νιώθει ότι είναι Ευρωπαίος και ακριβώς ε, να λάβουμε υπόψη μας τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις κοινέ απειλές, αλλά και τα περιβαλλοντικά ζητήματα της σήμερον ημέρα. Παρακαλώ να μιλάτε λίγο πιο αργά, λέει η Πρόεδρος, γιατί ναι, οι διερμηνείς υποφέρουν. Έλεγα λοιπόν ότι οι πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης είναι ο καλύτερος τρόπος για να νιώσει ο κόσμος ότι είναι Ευρωπαίοι και έτσι να αντιμετωπίσουμε από κοινού θέματα, απειλές, τα περιβαλλοντικά και να φτάσουμε στον κόσμο και μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας. Έπειτα, ε, diversity. Delta, diversity, D. Η ποικιλομορφία. Είναι πράγματι δύσκολο να το κατανοήσουμε αυτό. Έπειτα, ε για European Dimension. Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που διαφέρουν τους Ευρωπαίους σε εθνικό επίπεδο, σε τοπικό επίπεδο πρέπει να καταλάβουμε ότι το, η αίσθηση του ανήκειν δεν είναι κάτι καθαρά ευρωπαϊκό. F, funding, χρηματοδότηση. Οι πόλεις πιστεύουν ότι θα έχουν κάποιο οικονομικό κέρδος, ότι θα έχουν κάποια συνεισφορά. Και η Μελίνα Μαρκούρη το είπε αυτό στην αρχή με προπολογισμό που να βασίζεται σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Εγώ ζητάω το βραβείο Μελίνα Μερκούρη να αυξηθεί και η επιλογή μιας πόλης προκειμένου να είναι πολιτιστική πρωτεύουσα να είναι κάτι επιπλέον από τα άλλα προγράμματα. G για goal, στόχος. Ε, τι στόχο μπορούμε να μετρήσουμε και να κατανοήσουμε εσείς οι ευρωβουλευτές, τι στόχο έχετε για αυτά τα προγράμματα. Τι θέλουμε να πετύχουμε κάθε χρόνο. H, Human Rights, ανθρώπινα δικαιώματα. Αν δεν στηρίζει την οικουμενική δήλωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα μια πόλη, πιστεύω ότι δεν θα έπρεπε πότε να γίνει πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. I, impact. Θα πρέπει ο πολιτισμός να βάζει το μέτρο σε μια πόλη. Και αυτό από το 2030 η UNESCO ανακοινώνει δείκτες για αυτό το θέμα. Γιατί αν συνεχίσουμε να μετράμε την επιτυχία των πολιτιστικών πρωτευουσών βάσει της οικονομίας ή του τουρισμού, τότε δεν χρειαζόμαστε καλλιτέχνες, χρειαζόμαστε μόνο καλό μάρκετινγκ, διαφημίσεις, τίποτα άλλο. Κοιτάξτε, μιλάτε πάρα πολύ γρήγορα, λέει η Πρόεδρος, και όχι μόνο, ούτε και οι βουλευτές μετά δεν μπορούν να σας καταλάβουν. Όταν μιλάτε τόσο γρήγορα, σας δίνω δύο λεφτά παραπάνω για να περιορίσετε λίγο το ρυθμό σας, να μιλάτε λίγο πιο αργά. Α, ωραία, αυτό ήθελα να ακούσω, αυτό περίμενα, ευχαριστώ. Ωραία. J, jobs, απασχόληση. Τι κάνουμε με τις επιπλέον θέσεις απασχόλησης που δημιουργήθηκαν στις ευρωπαϊκές πολιτιστικές πρωτεύουσες. Ένα παράδειγμα είναι ότι μετά από το έτος που είναι μια πόλη πολιτιστική πρωτεύουσα υπάρχει ένας όρος κόσμος με υψηλά προσόντα που αναγκάζεται είτε να φύγει να πάει σε άλλη πόλη ή να βρει κάποια άλλη δουλειά χαμηλότερων προσόντων. Χρειαζόμαστε λοιπόν δίκτυα. Και είναι κάτι που το έχουμε πει ότι υπάρχει δίκτυο, αλλά δεν είναι ένα επίσημο δίκτυο, είναι μια οικογένεια, γιατί αγαπιόμαστε μεταξύ μας γιατί ε, συνεργαζόμαστε, περνάμε από τις ίδιες καταστάσεις, αλλά δεν πρόκειται για επίσημο δίκτυο. Τα πιο μακροχρόνια προγράμματα πολιτισμού στην Ευρώπη δεν γίνονται μέσω δικτύων. Είναι η πραγματικότητα, απλώς. Έπειτα, ε, know-how, γλώσσες, γλωσσικό. Εδώ πολλά μπορούμε να κάνουμε. Πρέπει να φροντίσουμε να διαχειριστούμε τα γλωσσικά δικαιώματα στην Ευρώπη και αυτό είναι μια πρόκληση. Μάρκετινγκ τώρα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να επενδύει πολύ περισσότερα χρήματα στην πρόθεση και την ε, διαφήμιση του τίτλου της πολιτιστικής πρωτεύουσα. Σίγουρα το γνωρίζετε ότι κάποιες ε, πόλεις, ωραία, γίνονται γνωστές, αλλά σε εσά. Όμως, εκτός από εσά ε, τα ξέρουν τα περί πολιτιστικών πρωτεύουσών, οι γειτονές σας, οι γονείς σας. Καμιά φορά συγκρίνουμε το θεσμό αυτόν με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δεν είναι όμως τόσο γνωστός. Είχαμε πολλές πρωτεύουσε και πόλεις στο πρόγραμμα, αλλά τελικά αυτοί που κερδίζουν είναι συνήθως πιο μικρές πόλεις που δεν έχουν προπολογισμό για να κάνουν ε, marketing όπως ήταν το Λίβερπουλ ή η Βαρκελόνη. Οπότε μη ζητάτε από μικρές άγνωστες πόλεις να πληρώσουν για αυτό τον τίτλο. Δικτύωση. Όπως είπα και πριν, χρειαζόμαστε μια πραγματική δικτύωση, ένα πραγματικό δίκαιο, ε, δίκτυο. Συγγνώμη. Πρέπει να είναι το μεγαλύτερο και το ισχυρότερο δίκτυο, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά κατά πάσα πιθανότητα και σε ολόκληρο τον κόσμο. Πόσες πόλεις, Oblivion, έτσι, πόσες πόλεις ξεχάστηκαν και ξέχασαν και οι ίδιες ότι κάποτε ήταν πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης σκεφτείτε, πηγαίνετε ε, στα, στις ιστοσελίδες των Δήμων και θα δείτε ότι δεν αναφέρεται τίποτα. Αυτό μας είναι αποτυχία. Πι, για πάρτι. Έχουμε πάρα πολλές ευκαιρίες που προσφέρουμε για γιορτές και όντω είναι μια ευκαιρία για γιορτή, για να συμβρεθούμε, γιατί είμαστε Ευρωπαίοι, γιατί έχουμε κοινέ αξίες, αλλά μπορούμε να περάσουμε μαζί και χρόνο. Q, για quality η καλλιτεχνική ποιότητα. Και αυτό είναι κάτι που βέβαια δεν φτάνουν 7 λεπτά για να το εξηγήσει κανείς, οπότε περνάω στο επόμενο, residencies. Η κάθε πόλη θα πρέπει να αποτελεί μέρος ενός ε, προγράμματος residence program στον κόσμο. Εγώ να σας πω ότι υπάρχουν 60 ε, πόλεις που το κάνουν αυτό. Τουρισμός. Έχω να ρωτήσω πόσοι από εσά έχετε πληρώσει από την τσέπη σα όταν πήγατε σε μια πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης πάνω από 300 χιλιόμετρα από την πόλη όπου μένετε. Αν δεν βρίσκεται στην κεντρική Ευρώπη, τότε πηγαίνουν μόνο πολίτες που ζουν στη γύρω περιοχή. Οπότε μην τους ζητάτε κάτι παραπάνω. Ε, ο θεσμός αυτός των πολιτιστικών πρωτεύουσων θα πρέπει να αποτελεί τη μέκα της Ευρώπης. Θα πρέπει να μπορούμε να προσαρμοστούμε στην κάθε περίπτωση. Αλλιώς είναι στην Ισπανία, στη χώρα των Βάσκων, που τον εθελοντισμό τον καταλαβαίνει κάποιο σαν τη δουλειά και είναι πολύ επικίνδυνο. Πρέπει λοιπόν να συμφωνηθεί. Έρχομαι στο W. Κάτι το οποίο έχω ήδη συζητήσει με κάποια μέλη της Επιτροπής αυτής όταν ήρθατε στο Σαν Σεμπαστιάν το 2016. Μετά από 35 χρόνια δεν νομίζετε ότι πρέπει να ξεκινήσετε να δημιουργείτε μία λευκή βίβλο για τις ευρωπαϊκές πολιτιστικές πρωτεύουσε, τη βίβλο της πολιτιστικής Ευρώπης που δεν έχει γραφτεί ακόμα. Αλλά όχι να τη γράψετε και να τη φωτοτυπήσετε και τελείωσε μην την ξεχάσετε και μην ξεχνάτε τι έχουν κάνει προηγούμενοι να προσαρμοζόμαστε από κάτω προς τα πάνω και από πάνω προς τα κάτω. Και έρχομαι στο τέλος year, έτος, πέντε χρόνια. Μήπως θα έπρεπε να γίνουν τρία, να δηλαδή προσαρμόσουμε το πρόγραμμα και να έχουμε κάθε τρία χρόνια. Το 2017 ήταν που μπήκανε κριτήρια μέχρι το 2033. Δεν θα έπρεπε να αλλάξει αυτό. Γιατί αλλιώς τα τελευταία χρόνια, τελευταίες δηλαδή πολιτιστικές προτάσεις ε, δεν θα είναι πια προσαρμοσμένες στην πραγματικότητα. Δυστυχώς η πραγματικότητα προχωράει πιο γρήγορα από αυτό το πρόγραμμα. Και έρχομαι στο τελευταίο γράμμα Z. Γιατί οι βόρειες και οι δυτικές ε, χώρες δεν είναι τόσο πρόθυσμες να είναι υποψήφιες οι μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις έχουν πολλά να θυμούνται και έχουν πολλά να θυμούνται από το παρελθόν τους. Αυτό είναι ένας λόγος. Το δεύτερο είναι ότι δεν υπάρχει καλή προσαρμογή και ακόμα προσπαθούμε να βρούμε τον κατάλληλο ρυθμό. Η Δυτική Ευρώπη κοιτάζει το θεσμό αυτό σαν κάτι παλιό από το παρελθόν, ενώ η Ανατολική Ευρώπη βλέπει το θεσμό σαν κάτι στο οποίο προσβλέπει. Αυτά από το Α μέχρι το Ζ και ζητώ συγγνώμη από τους διερμηνείς, λέει ο μιλητής. Thank you very much Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την ε, πολύ καλά δομημένη και ε, πολύ εμπεριστατωμένη παρουσίαση. Θα ήθελα τώρα να δώσω τον λόγο στον Γύρι Σουτσάνεκ, ε, πρώην CEO της πολιτιστικής πρωτεύουσας ε, του Πίλσεν για το 2015. Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Εγώ αποφάσισα, μια και κοντεύουν Χριστούγεννα, να ε, είμαι λίγο πιο νοσταλγικός. Και ε, του χρόνου θα είναι άλλωστε και η πέμπτη επέτειος μετά την πολιτιστική πρωτεύουσα του Πίλσεν και θα ήθελα να σας δείξω κάποια στοιχεία τα οποία ήταν επιτυχία και άλλα τα οποία αποτέλεσαν δική μας αποτυχία ή μάλλον δική μου αποτυχία. Είχαμε ένα τουριστικό, μια τουριστική κίνηση πολύ σημαντική. Ε, πρέπει να πω βέβαια ότι αποτέλεσε η πολιτιστική πρωτεύουσα το πιο μεγάλο ε, πολιτιστικό ε, γεγονός στην τσεχική δημοκρατία με προϋπολογισμό περίπου 68 εκατομμύρια, 18,2 όσον αφορά μη δαπάνες υποδομής και τα υπόλοιπα για τις δαπάνες υποδομής. Εγώ θα ήθελα να μιλήσω για τις αλλαγές που έγιναν στην διαχείριση, γιατί συχνά συμβαίνει αυτό και αυτό προκαλεί πολύ συχνά επίσης δυσκολίες. Και ε, να ε, μιλήσω και για την ισορροπία που ανέφερε προηγουμένως ο Ξάβη, ε, γιατί πρέπει να υπάρχει όντως ισορροπία μεταξύ όλων των στοιχείων. Ισορροπία. Λοιπόν, εδώ βλέπετε σε κόκκινο την πολύ χαμηλή συμβολή της εθνικής κυβέρνησης. Όπως είπε και ο Ξάβη, ε, θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει. Αξίζει ο θεσμός για περισσότερη συμβολή ε, και κάποιες χώρες ε, θα πρέπει να σκεφτούν ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν την δυνατότητα να συμβάλλουν περισσότερο Πάντως, ε, οτιδήποτε μας υποσχέθηκαν, μας το έδωσαν. Οτιδήποτε υποσχεθήκαμε εμείς ότι θα κάνουμε, το κάναμε και ε, τα χρήματα βγήκαν από τον κοινοτικό προϋπολογισμό, δηλαδή της πόλης, του Δήμου. Ε, εδώ βλέπετε ένα θαυμάσιο νέο θέατρο, το οποίο χτίστηκε ε, χάρη του προγράμματος και αποτελεί ακόμα μία από, τις, από τα σημαντικά σημεία επίσκεψης και ενδιαφέροντος στην πόλη μας. Εδώ βλέπετε δύο κόκκινες γραμμές, 42 περίπου εκατομμύρια ευρώ, μας κόστησε το νέο θέατρο ε, και περίπου 500.000, δηλαδή μισό εκατομμύριο, ε, εκατομμύρια, ε, η ζώνη η οποία έγινε πολύ γνωστή το ΝΤΕΠΟ 2015. Εάν φανταστείτε πόσα προγράμματα έγιναν σε αυτό το νέο θέατρο, λίγα γιατί δεν υπήρχε ε, ε, προετοιμασία και επομένως χτίστηκε πραγματικά την τελευταία στιγμή ε, και επομένως δεν ήταν έτοιμο έγκαιρα το θέατρο. Ωστόσο τώρα έχουμε πλέον το θέατρο αυτό, είναι επιτυχημένο και ε, γίνονται εκδηλώσεις και τα λοιπά, αλλά ξέρετε καμιά φορά τα legacy programs, αυτά δηλαδή που ε, εντυπώνονται ε, και χτίζονται με την πόλη, μπορεί να είναι μερικά πολύ μικρότερα, έως και πολύ μικρά. Πολλές χώρες είχαν άμεση ανάμειξη με τα projects, έγιναν συνεργασίες με την Γερμανία, με την Ιαπωνία, με τη Γαλλία και με άλλες χώρες. Αυτό ε, σημαίνει ότι αν θέλετε πραγματικά να δημιουργήσετε κληροδότημα, αν θέλετε legacy, ε, θα πρέπει να δαπανηθούν κάποια χρήματα. Φυσικά υπάρχουν και αυτά τα πολύ όμορφα προγράμματα, ε, εκατοχιλιάδες άνθρωποι το είδαν και πραγματικά ήταν περηφάνεια για τους ντόπιου ε, Πολωνοί, Τσέχοι και άλλοι καλλιτέχνες επίσης συμμετείχαν σε αυτό. Επίσης έχουμε εδώ ε, επίδραση πάνω σε πιο καινοτόμα προγράμματα, ακόμα και σε παρεμβάσεις που αφορούν αρχιτεκτονικά ε, στοιχεία της πόλης Οπωσδήποτε όμως και ε, το τονίζω αυτό και ο Δήμος και η Περιφέρεια ε, θα πρέπει να βοηθήσουν. Εδώ έχουμε μια μεγάλη παραγωγή από την Περιφέρεια τους κατοίκους ε, του Πίλσεν και ήταν ένα από τα πιο συγκινητικά προγράμματα και συγκινητικές στιγμές ε, όλου του προγράμματος. Έρχομαι εδώ ε, στο κύριο ε, πρόβλημα ή την, την κύρια πρόκληση που είναι το κληροδότημα. Τι μένει το να, είναι, να γίνει ένα διεθνές μπραντ, να δημιουργηθούν νέε υποδομές, να δημιουργηθούν δίκτυα προγραμμάτων πολιτιστικού χαρακτήρα, καθώς επίσης και στοιχεία της δημιουργικής της βιομηχανίας. Ε, ε, ε, χαιρόμαστε πάρα πολύ γιατί τα τα μία έχουν ταμεία έχουν μια νέα περίοδο και αυτό είναι πολύ καλό. Όσον αφορά το Legacy Projects, εδώ βλέπετε ένα κέντρο συγκεκριμένο στο PILS, είναι και χώρος παρουσίασης εκδηλώσεων, αλλά είναι και χώρος όπου πολλά προγράμματα διεθνούς συνεργασίας ε, έλαβαν ε, χώρα. Έχουμε οργανώσει ας πούμε το φεστιβάλ Μπαρόκ, έχουμε ε, οργανώσει επίσης τη σειρά εκδηλώσεων Μπαβάρια κλπ. Πρόκειται για ένα κτίριο το οποίο χρησιμοποιήθηκε πολύ και ακόμα το χρησιμοποιούμε. Δημιουργήσαμε επίσης ένα φεστιβάλ με φώτα ε, που λέγεται Blick μπλικ καταφέραμε να φέρουμε από όλα τα μέρη της χώρας αλλά και από διαφορετικές χώρες ανθρώπους με διαφορετικό υπόβαθρο ε, και ε, νομίζω ότι και η Ιάννα θα σας πει μετά για την Ρίγα γιατί χρησιμοποιήθηκαν τα ίδια στοιχεία κάποια άλλα legacy projects έχω βάλει εδώ για την περίπτωση του Πίλσε. Είχαμε ας πούμε και μικρά, μικρής εμβέλειας γεγονότα όπως η ημέρα, η Ευρωπαϊκή ημέρα των γειτόνων. Ε, αναφέρθηκα προηγουμένως στο Baroque Festival ε, Τσεχίας και Βαβαρίας. Ε, έχουμε κι άλλα ε, και οπωσδήποτε ε, βλέπουμε και διάφορα στοιχεία τα οποία αφορούν τον εθελοντισμό πάντα μέσα στη δημιουργική βιομηχανία και μια σειρά από άλλα προγράμματα τα οποία αφορούσαν την πρωτεύουσα. Αυτή είναι η ιστορία του Πίλσεν. Εγώ ε, εξακολουθώ να εκπροσωπώ την πόλη και τις δραστηριότητες ε, του κληροδοτήματος, αυτά που εμείς ονομάζουμε legacy activities, ε, αλλά ξέρετε πρόκειται για εύθραυστη κατάσταση. stay in the city and uh, the organization team needs to take it in mind from the very beginning. Ε, γιατί πρόκειται για ε, θέματα τα οποία συνήθως τα κουβαλάνε αν θέλετε και τα προωθούν πολύ μικρός αριθμός ατόμων. Γι' αυτό είναι δύσκολο. Αυτά είχα να σας πω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Τελευταίος ομιλητής ε, στον πρώτο γύρο πριν ξεκινήσουν οι ερωτήσεις είναι ο Ταμάς Ζαλάη σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ αποφάσισα να, ε, να τιμήσω την ε, ποικιλία. Γι' αυτό λοιπόν θα μιλήσω ούτε ογκρικά, ούτε αγγλικά, αλλά θα μιλήσω γερμανικά. Ε, πάρα πολύ σύντομα να σας παρουσιάσω το τι έγινε τότε στο pitch. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι μπορούμε να αναγνωρίζουμε τα λάθη μας. Ε, πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί, αυτό ήδη ελέγχθη και επιτρέψτε να φέρω και ε, κάποια ιστορία. Το δικό μας, η πόλη μας ήταν το Πέτσο το 2010, ε, πολιτιστική πρωτεύουσα με την πόλη Έσεν και την Κωνσταντινούπολη. Ξεκινήσαμε ήδη το 2004. Το 2004 ήταν ε, μια πολύ ενδιαφέρουσα χρονιά στην Ουγγαρία, γιατί τότε προσχωρήσαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν λοιπόν ένα νέο ξεκίνημα αλλά βεβαίως υπήρχαν τότε και πάρα πολλές δυσκολίες και θα σας εξηγήσω πολύ σύντομα ποιες ήταν αυτές. Ε, όσον αφορά το πλαίσιο, ε, όπως ε, σας είπα, ξεκινήσαμε τις ε, προετοιμασίες το 2004 και ε, εκεί προέκυψε μια σημαντική αλλαγή, δηλαδή μεταξύ του 2085 και του 2091 κατ' ουσίαν ε, εορτάσαμε τον μεγάλο ε, ευρωπαϊκό πολιτισμό. Και το 1991 στην Μέση διάταξη των πολιτιστικών πρωτευουσών στην ημερήσια διάταξη τέθη το θέμα της ανάπτυξης της πόλης, της δυνατότητας μιας πόλης να εξελιχθεί περαιτέρω. Αυτό λοιπόν μας ενέπνευσε και τότε αποφασίσαμε και εμείς ε, να συμμετάσχουμε με 10 περαιτέρω πόλεις ε, στην Ουγγαρία. Ήμασταν λοιπόν 11 υποψήφιες πόλεις και είχαμε, επιλέξαμε τρία μεγάλα θέματα. Ε, θέλαμε να εκδημοκρατικοποιήσουμε την έννοια του πολιτισμού. Δηλαδή, ε, πώς μπορεί κανείς ε, να διαμορφώσει πολιτισμό με συμμετοχή δική του, να έχει δημοκρατικές δομές. Αυτό ήταν ε, ένας πολύ σημαντικός στόχος. Ένας άλλος στόχος ήταν ότι δώσαμε ιδιαίτερη σημασία στο διαπολιτισμικό στοιχείο. Είπαμε ότι αυτό είναι αξία. Θα την εορτάσουμε ε, και θα την ε, βραβεύσουμε ως αξία και λόγω της, ε, των πολλών εθνοτήτων θέλουμε να είμαστε πιο διεθνιστές, δηλαδή αυτό το διεθνιστικό στοιχείο να το εκμεταλλευτούμε ως μια πηγή έμπνευσης. Αποφασίσαμε λοιπόν να προβάλλουμε περισσότερο τις οικαστικές τέχνες και όχι μόνο τα φολκλωρικά στοιχεία. Το τρίτο που θέλω να πω ήταν ε, μετά την αλλαγή στο Λέσκου και εμείς ε, πιστεύαμε ότι το ΠΕΤΣ, η δική μας ήταν σε μια μεταβιομηχανική φάση και θέλαμε τη βιομηχανία που χάθηκε να την αντικαταστήσουμε με πολιτισμό, να ενισχύσουμε την πόλη πολιτιστικά. Αυτοί ήταν οι τρεις βασικοί μας στόχοι και βεβαίως είχαμε να αντιμετωπίσουμε και προκλήσεις. Μερικές προκλήσεις ήταν πολύ μεγάλες και δεν μπορούσαμε να τις ξεπεράσουμε. Το 2004 είχαμε ακόμα τις παλιές κομμουνιστικές δομές που ήταν έντονα παρούσες, αυτή την οτροπία από πάνω προς τα κάτω και αυτό θέλαμε να το χαλαρώσουμε και στο, στους πολιτικούς και ε, σε επίπεδο πολιτών. Η Ουγγαρία είναι ακραία συγκεντρωτικό κράτος. Όλα γίνονται στη Βουδαπέστη οτιδήποτε γίνεται εκτός Βουδαπέστης είναι αόρατο. Δεν το λαμβάνει κανείς υπόψη του. Εμείς λοιπόν θέλαμε να επιδιώξουμε την αποκέντρωση και αυτό δεν ήταν απλό. Ε, το 2004 με την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, κληθήκαμε να εναρμονίσουμε και την νομοθεσία μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό συνεπάγει συνεπάγεται μεγάλα προβλήματα, κυρίως στο σχεδιασμό. Οι νόμοι για τους δημόσιους διαγωνισμούς, για την προκήρυξη αυτών των διαγωνισμών, ε, άλλαζαν συνεχώς και χρειάστηκε να περάσει κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι να αποκτήσουμε μια ουσιαστική νομική βάση. Ε, νομίζω ελέγχθη προηγουμένως ότι αυτό που ενδιέφερε ιδιαίτερα ήταν η ματιά της Ανατολικής Ευρώπης. Από τις Βρυξέλλες αυτό δεν ήταν ιδιαίτερα συνειδητό, αλλά παρόλα αυτά εμείς ε, συνειδητοποίησαμε ότι χρειαζόμαστε κατ' ουσίαν ένα κοινό λεξικό. Γιατί, Γιατί λέγαμε, χρησιμοποιήσαμε τις ίδιες λέξεις, αλλά οι λέξεις αυτές σημαίνουν κάτι τελείως διαφορετικό ε, στη Δυτική Ευρώπη από ότι στην Ανατολική Ευρώπη. Και δεν είναι ότι δεν είχαμε εμείς ε, κανόνες για τους ε, διαγωνισμούς. Είχαμε, ε, βέβαια όλα αυτά δεν ήταν τόσο απλά. Αναγκαστήκαμε να δημιουργήσουμε ένα άτυπο δίκτυο πολιτιστικών πρωτοβουσών. Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, χρειαζόμαστε μία πλατφόρμα για ανταλλαγές, για capacity building, για ανταλλαγή εμπειριών. Αποτέλεσμα όλων αυτών με την πρώτη ε, στοχοθέτησή μας που ήταν όπως σας είπα να εκδημοκρατικοποιήσουμε τον πολιτισμό. Αυτό για μας ε, ήταν ένα πολύ μεγάλο λάθος γιατί δεν το καταφέραμε. Ήταν ένα πολύ μεγάλο καθήκον αυτό που αναλάβαμε και κατ' ουσίαν αυτό ήταν η πιο μεγάλη σκιά που έπεσε τότε στο ΠΕΤΣ. όσον αφορά την διαπολιτισμική ε, περιφέρεια, αυτό είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα κληρονομιά με τους ε, Κροάτες και τους ε, Σέρβους, τη μειονότητα στο πιτς, τη μειονότητα αυτών των δύο εθνοτήτων. Ξεκινήσαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνεργασία. Εξακολουθούν να υπάρχουν κάποια στοιχεία αυτής της συνεργασίας ακόμα και σήμερα. Και αυτό που έχει σημασία είναι ότι το πιτς είναι πλέον ορατό ως ένας διεθνής χώρος. Επιπλέον, ε, ένα εργοστάσιο κεραμικών το μετατρέψαμε σε πολιτιστικό κέντρο. Αυτό δεν ήταν καθόλου εύκολο, ε, γιατί δεν ενδιέφερε κατ' ουσίαν κανένα στη χώρα. Αυτό που ενδιέφερε ήταν μόνο αν ήταν έτοιμες ε, οι υποδομές. Άρα δηλαδή είχαμε να αντιμετωπίσουμε πολλές δυσκολίες κατά τη φάση της εφαρμογής, αλλά πρέπει να σας πω ότι αυτή είναι η πιο σημαντική κληρονομιά που έμεινε στην πόλη. Η πόλη έχει αλλάξει, μπορώ να σας δείξω φωτογραφίες, αλλάξαμε ε, τα πάρκα, ε, αλλάξαμε έναν δρόμο που οδηγεί στο μουσείο, φτιάξαμε μια νέα βιβλιοθήκη. Όπως ε, σας είπα, αυτό το εργοστάσιο κεραμικών το μετατρέψαμε σε πολιτιστικό κέντρο και φτιάξαμε επίσης ε, και μία αίθουσα για συναυλίες. Ε, με τη σημερινή μου εμπειρία θεωρώ ότι αν θέλει κανείς ε, να έχει μία πόλη πλούσια σε πολιτισμό, τότε είναι πολύ σημαντικό να αντιμετωπίσει κανείς τα προβλήματα. Τα πολιτιστικά, τα αστικά, να φτιάξει ένα σχέδιο για το πώς μπορούν να ξεπεραστούν τα προβλήματα αυτά. Και αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι όλα αυτά ε, θα πρέπει να γίνονται με ουσιαστική συμμετοχή στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Και το τελευταίο που θέλω να πω, η τελευταία μου πρόταση είναι, ε, κατά την άποψή μου, υπάρχει ένα θέμα όπου οι πόλεις ε, χρειάζονται ακόμα βοήθεια από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό είναι η πολιτική επιρροή. Ε, δηλαδή για τις ε, πόλεις που έχουν ήδη ανακηρυχθεί ως πολιτιστικές πρωτεύουσες και τα πράγματα είναι καλύτερα για τις υποψήφιες πόλεις δυστυχώς δεν προκύπτει ουσιαστική υποστήριξη γιατί εμφανίζονται νέες ομάδες που θέλουν την υποστήριξη των πολιτικών. Εγώ ε, σε αυτό θα περίμενα κάποια μεγαλύτερη υποστήριξη από τις Βρυξέλλες. Σας ευχαριστώ. Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι αυτά που ακούσαμε ήταν όλα πολύ ενδιαφέροντα. Ε, το να ακούσουμε ε, μια άποψη από την εμπειρία, το τι πρέπει να γίνει και τι δεν πρέπει να γίνει και ε, θα ήθελα τώρα ε, να δώσω τη δυνατότητα ε, στους συμμετέχοντες να θέσουν ερωτήσεις. Δεν ξέρω, έχετε ερωτήσεις. Η Πέτρα, Κάμα Εύερτ και μετά θα ακολουθήσουν και άλλοι. Thank for... Ευχαριστώ πολύ, λέει κυρία Σέντροβα για, την, ε, για τις παρουσιάσεις σας, ε, για όσα είπατε και για τον ενθουσιασμό σας. Γιατί ξέρουμε ότι κάνετε μεγάλες προσπάθειες για τις δραστηριότητες αυτές των ευρωπαϊκών ε, πολιτιστικών πρωτεύουσών. Έχω δύο ερωτήσεις. Είπατε ότι υπάρχει ανάγκη για πολιτική στήριξη. Για σας συγκεκριμένα, στη δικιά σας την πόλη, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων, Υπάρχει, υπήρξε αρκετή στήριξη, γιατί στο Πίλσεν ξέρουμε ότι δεν ήταν τόσο εύκολα τα πράγματα. Υπήρξαν ε, αλλαγές στην πολιτική εκπροσώπηση. Φαντάζομαι και στις τρεις πόλεις υπάρχει το ζήτημα αυτό. Είναι, πώς να το πω, δύσκολο να συνεχίζουμε και να εξηγούμε και να πείθουμε τον κόσμο για το πόσο μεγάλη σημασία έχει το πρόγραμμά σας και σίγουρα ακόμα περισσότερο αν δεν υπάρχει πολιτική στήριξη. Δεύτερη ερώτηση. Από ό,τι πετύχατε, η πόλη σας έγινε πιο γνωστή στην Ευρώπη. Εγώ πιστεύω πως ναι, αυτό είναι σίγουρο. Όμως, στην πόλη σας. Τώρα ο θεσμός είναι πιο γνωστός. Από ότι γενικότερα έχετε γνώμη από αυτού. Κοιτάξτε, ε, καλύτερα να συγκεντρώσουμε κάποιες ερωτήσεις, ε, να τις ομαδοποιήσουμε ανά τρεις. Ε, θα απαντάτε και μετά άλλες πάλι τρεις, καλύτερα έτσι. Η Πέτρα λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ και για τις πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσει. Εγώ έχω μία πολύ απλή ερώτηση που βέβαια φοβάμαι ότι θα είναι δύσκολο να απαντηθεί. Δηλαδή όταν κάποια στιγμή την προτελευταία θητεία δώσαμε νέο προσανατολισμό στις πολιτιστικές πρωτεύουσες, κρίναμε τότε ότι δεν θα πρέπει να είναι ένα γεγονός για ένα μόνο χρόνο, αλλά να υπάρχει κάποια βιωσιμότητα. Δηλαδή, μετά από αυτό το χρόνο όπου θα έχουμε ωραίες γιορτές, σημαντικό αυτό, μετά όμως να παραμένει κάτι στις ε, πόλεις και να υπάρχει και μία βιώσιμη εξέλιξη στην πόλη. Γι' αυτό λοιπόν απλή αλλά πολύ σημαντική ερώτηση. Τελικά τι σας έμεινε από αυτή τη διαδικασία. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πολύ για τις παρουσιάσεις σας. Θέλω να ρωτήσω τον Χαβιέ και να προφέρω σωστά το όνομά σας. Βρήκα πολύ ενδιαφέροντα τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάσατε τα διάφορα σημεία που είχατε να μας παρουσιάσετε για τις πολιτιστικές πρωτεύουσες εκφράσατε κάποιες αμφιβολίες για τον πενταετή ρυθμό της διαδικασίας. Εγώ όμως θέλω να εκφράσω τις αμφιβολίες μου γι' αυτό. Κυρίως αν λάβουμε υπόψη μας ότι μπορεί να υποφεληθεί ο πολιτιστικός ο κλάδος από τις υποδομές. Αν ήταν τρία χρόνια δεν θα ήταν το ίδιο. Μπορείτε να μας δώσετε λοιπόν τα δικά σας επιχειρήματα. Επίσης, Θα ήθελα να ακούσω και από τους άλλους να εξηγήσουν τη θέση τους από αυτού. Ωραία, να δώσουμε το λόγο στους εμπειρογνωμονές μας εδώ για να απαντήσουν σε αυτές τις πρώτες ερωτήσεις, παρακαλώ. Ωραία, θα μιλήσω ισπανικά αυτή τη φορά. Πρώτα απ' όλα, για τα θέματα που έχουν να κάνουν με την πολιτική στήριξη. Το Σαν Σεμπαστιάν καθ' όλη την διαδικασία είχε συνέχεια αλλαγέ. Κάθε φορά που είχαμε εκλογέ υπήρχαν αλλαγέ, για να το πω έτσι σύντομα. Οπότε, σε όλε τι περιπτώσει, η στήριξη των πολιτικών ήταν απόλυτη. Αλλά όταν αλλάζει ένας πολιτικός, αλλάζει και το όραμα. Έχουμε εκλογές, οπότε ξέρετε, εσείς ε, μπορεί να θέλετε όλοι να στηρίξετε τον πολιτισμό, αλλά τον βλέπετε διαφορετικά. Οπότε, για να σας απαντήσω, αυτό που είναι ζωτική σημασία για μένα είναι το διευθυντικό όργανο δεν θα έπρεπε να έχει πολιτικοποιηθεί τόσο. Θα έπρεπε να έχει μεγαλύτερο βάρος πολιτιστικό, κοινωνικό. Αυτό θα ήταν το καλό και δεν το λέω μόνο εγώ αυτό. Σε αντίστοιχες περιπτώσεις και άλλοι που παρακολούθησαν την κατάσταση τα ίδια είπαν. Πιστεύω ότι είναι ζωτική σημασία σε αυτό. Δεύτερον, κατά πόσο ε, η Ευρώπη είναι περισσότερο ορατή στο Σαν Σεμπαστιάν από ό,τι κατά το παρελθόν. Ναι, σίγουρα, αλλά τι ήταν η Ευρώπη, ήταν συμμεταχή, ήταν συνεργασία, ήταν προγράμματα, ήταν να ανακαλύψουμε το πολωνικό θέατρο, ήταν να ανακαλύψουμε άλλες χώρες και ένα σωρό ανθρώπους, καλλιτέχνες κλπ. Γιατί αν χρειαζόμαστε κάτι ακόμα στην Ευρώπη, αυτό είναι διαπαιδαγώγηση. Θα έπρεπε να γνωριστούμε, να καταλάβουμε ο ένας τον άλλον. Πρώτα απ' όλα πρέπει να δώσουμε τα χέρια μεταξύ μας. Βλέπετε, έχω τέτοιο πάθος όταν μιλάω για αυτά που δεν κρατιέμαι. Δεύτερο σχόλιο τώρα. Λέτε, τι έμεινε. Η κληρονομιά. Λοιπόν, ναι. Τώρα τελειώνει ε, η περίοδος του 2007-2009 που έβαζε συγκεκριμένα κριτήρια για την κληρονομιά. Τώρα περνάμε στην τρίτη περίοδο, 2021 ε, με 33. Αυτό που θα έλεγα λοιπόν είναι ότι στο προηγούμενο τουλάχιστον ψήφισμα πάντα υπήρχε δυνατότητα 31 Δεκεμβρίου, όπως λέει και ένας εμπειρογνώμονας ο Steve Green, η ευρωπαϊκές πολιτιστικές πρωτεύουσε μπορούν να σβήσουν το φως και να κλείσουν την πόρτα. Κάτι το οποίο όμω δεν θα έπρεπε να συμβεί ποτέ. Εάν μια πόλη θέλει να υποβάλει υποψηφιότητα, είναι γιατί θέλει να αποτελέσει μέρος της οικογένειας για πάντα, χωρίς αυτό να σταματήσει ποτέ. Και για τις ερωτήσεις σας όσον αφορά τα πέντε χρόνια και τη Λευκή Βίβλο, στην περίπτωση των πέντε ετών η απάντηση για τις υποδομές είναι κάτι που εύκολα λύνεται, γιατί οι υποδομές δεν προσαρμόζονται στα πέντε χρόνια. Έχουμε παραδείγματα πρωτευουσών που έχουν σταθμούς που δεν έχουν ολοκληρωθεί τρένων, ας πούμε, ή λεωφορείων ή θέατρα που πήγανε, φτάσανε εκεί πριν. Θα συμφωνήσετε λοιπόν μαζί μου ότι δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στους επικεφαλείς των έργων, τους αρχιτέκτονες, τους κλπ, να αποφασίζουν πότε θα ολοκληρώνεται κάτι. Γιατί προτείνω τρία χρόνια, γιατί πιστεύω ότι όλα προσαρμόζονται. Και μία προσαρμογή όπου τον πρώτο χρόνο αποφασίζεται η πρωτεύουσα, έχει ένα χρόνο για να ολοκληρώσει το πρόγραμμά της η πόλη. Κάποιος που έχει τρία χρόνια ξέρει ότι έχει τρία, δεν έχει παραπάνω. Οπότε έτσι ξέρει ότι σε τρία χρόνια μπορεί να κάνει ό,τι έχει να κάνει και capacity building και εκπαίδευση του κόσμου και επικοινωνία. Ε, παραγωγή θα είναι μια κατάσταση καλύτερα προσαρμοσμένη στην πραγματικότητα, γιατί μιλάμε για πόλεις που κατά πάσα πιθανότητα προηγουμένω δεν ξέρατε καν που βρίσκονται στο χάρτη πριν γίνουν πολιτιστικέ πρωτεύουσε. Σε όλου μα συμβαίνει αυτό. Λοιπόν, αυτή είναι μια πραγματικότητα. Ζητάμε λοιπόν από αυτή την πόλη ξαφνικά να κάνει μια σούπερ παραγωγή. Νομίζω ότι τα τρία χρόνια είναι η κατάλληλη περίοδο και η Λευκή Βίβλος, το επαναλαμβάνω, για μένα θα ήταν τόσο εύκολο, τόσο απλό, σαν να συνοψίζαμε έναν οδηγό όπου θα λαμβάνονται υπόψη πάρα πολλά πράγματα για να προετοιμαστούμε. Σίγουρα χρειάζεται διαπαιδαγώγηση, αλλά θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Όλοι εδώ μπορούμε να μιλάμε για αλλαγέ στην ηγεσία όσον αφορά τη διαχείριση, για συγκρούσεις, γιατί όλοι περάσαμε από αυτά. Και τι γίνεται, όταν μας συμβαίνουν αυτά, σκεφτόμαστε ότι είναι η χειρότερη στιγμή του κόσμου και ότι είμαστε η χειρότερη ευρωπαϊκή πολιτιστική πρωτεύουσα του κόσμου. Το Πίλσεν, το Πέτσι, η Ματέρα, σε ολόκληρη την Ευρώπη να ξέρετε, δεν έχουμε ούτε μία περίπτωση ευρωπαϊκή πολιτιστική πρωτεύουσα που να κρατάει τη διεύθυνση από την αρχή μέχρι το τέλο. Αλλιώ, αν υπάρχει, εγώ να φτιάξω άγαλμα σε αυτή την περίπτωση, σε αυτό το άτομο που κατάφερε και βρέθηκε επικεφαλή από την αρχή μέχρι το τέλο. Πάντα υπάρχουν αλλαγέ. Οπότε, εγώ το είπα. Ε, λευκή βίβλος, αλλά χωρίς αυτό να σημαίνει να κάνουμε αντίγραφο. Όχι σημαίνει να έχουμε μια κατευθυντήρια γραμμή, ένα σημείο κίνησης αν με τι άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και κυρίω να ευχαριστώ του και τι διερμηνεί, ε, γιατί σήμερα πραγματικά η δουλειά του είναι κόλαση. Για και μιλάμε για πολιτικούς και πολιτική υποστήριξη, ε, θα μπορούσα να πω ότι ε, θα μπορούσα να μιλάω για δύο ώρες, αλλά εν πάση περιπτώσει να σας πω ότι είναι δύο ειδών τα προβλήματα. Είναι η έλλειψη υποστήριξη σε τοπικό επίπεδο πρώτα, που προκαλεί προβλήματα στην διάρθρωση, στην διαχείριση των προβλημάτων. Δεν ακολουθείτε το βιβλίο της προκήρυξης ε, και η συγγραφή υποχρεώσεων κτλ. Σε πολλές περιπτώσεις ε, προσπαθούμε να λύσουμε τα προβλήματα αυτά μέσα από αλλαγές στην ε, δομή της διαχείρισης. Το άλλο επίπεδο είναι το εθνικό. Εδώ ε, μπορεί να προκύψουν σημαντικά προβλήματα δυσχέρειες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Ας πούμε, υπάρχει μια χώρα, μια πόλη που έχει τον τίτλο για ε, το 2021 και παίρνει λιγότερο από το 20% του προϋπολογισμού που είχε υποσχεθεί η εθνική κυβέρνηση. Ε, μα αυτό σημαίνει ότι η Οργανωτική Επιτροπή στην πόλη αυτή θα έχει και έχει αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα. Εγώ θα έκανα ένα κανόνα που λέει ότι όταν εμπλέκεται η χώρα, η εθνική κυβέρνηση θα πρέπει να εκδώσει συγκεκριμένη επίσημη δήλωση σχετικά με το ύψος της συνεισφοράς έτσι ώστε να ξέρει η πόλη από την αρχή ότι θα έχει στη διάθεσή της ε, αυτά τα ε, χρήματα. Άσχετα εάν η πόλη διοικείται από φύλλα προσκύμενη κυβέρνηση, ε, συγγνώμη, φύλλα προσκύμενου στην κυβέρνηση ή είναι αντίθετη προς την κυβέρνηση. Ε, όσον αφορά τη δική μας περίπτωση, ναι, βεβαίως έχει γίνει πολύ πιο ορατή η ε, πόλη και η Ευρώπη είναι πιο ορατή. Ε, με τον τρόπο αυτό γίναμε μία από τις πιο φιλοευρωπαϊκές πόλεις ε, και νομίζω ότι πλέον έρχεται πολύ πιο φυσικά να πει κανείς να είμαι Ευρωπαίος και σε σχέση με το τι μένει έκανε στο Πλόβλιχ ε, ε, μία παρουσίαση σχετικά με το κληροδότημα που μας έχουν αφήσει. Μία ώρα μίλησα, δεν ήταν και τόσο εύκολο. Υπάρχουν όμως πολλά παραδείγματα ε, για τον τρόπο με τον οποίο ωφελήθηκαν, εποφελήθηκαν οι πόλεις από τον θεσμό της πολιτιστικής πρωτεύουσας. Ε, και ε, βεβαίως ξεκινούν ενδεχομένως ε, και μεγάλες εκδηλώσεις όπως είναι η Μπερλινάρε ή το ο διαγωνισμός κινηματογράφου του Βερολίνου και νομίζω ότι είναι και αυτά τρόποι μέσω των οποίων μπορεί να διατηρηθεί ε, το, κληροδόκημα, ε, το κληροδότημα, τρόποι με τους οποίους μπορεί κανείς ε, να διαχύσει κατά κάποιο τρόπο τα όσα έγιναν στην πόλη κατά τη διάρκεια της πολιτιστικής πρωτεύουσας. Και βέβαια μετά την προετοιμασία, την ίδια τη χρονιά της πολιτιστικής πρωτεύουσας, Ε, γίνεται η πολύ σοβαρή δουλειά και εγώ θα έλεγα ότι πάνω από το 50% των πόλεων παίρνουν πολύ σοβαρά αυτό τον τίτλο της πολιτιστικής Σε Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ζαλάη. Θέλω να σας πω ότι ε, δεν είμαι καθόλου τώρα σίγουρος αν μπορούμε να αρχίσουμε διάλογο, αλλά ξέρεις, ε, παρόλα αυτά, αυτό που πρότεινες, το να δεσμεύονται οι εθνικές κυβερνήσεις. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο και επικοδομητικό. Από την άλλη βέβαια μπορεί να είναι και αντιπαραγωγικό. Γιατί είμαι πεπισμένος ότι τελικά αν ε, οι κυβερνήσεις ε, δίδουν πολλά περισσότερα χρήματα από τις πόλεις, τότε μετατοπίζονται οι σχέσεις και αυτό εμείς το ζήσαμε στο πίτσε. Η πολιτική υποστήριξη είχαμε καθ' όλη τη διάρκεια της υποψηφιότητάς μας. Ε, οι πολιτικοί δεν ήθελαν να τους ενοχλούμε καθόλου. Λέγανε κάντε ό,τι θέλετε, σίγουρα θα είναι καλό το πρόγραμμα. Και όταν ανακηρυχθήκαμε πολιτιστική πρωτεύουσα, τότε οι πολιτικοί μας έδωσαν τη στεναρή υποστήριξή τους, διότι όπως σας είπα, ε, πλέον ε, είχε στραφεί το ενδιαφέρον ε, στις υποδομές μας. Και το 2010 ήταν έτος εκλογών στην Ουγγαρία, τόσο δημοτικών όσο και βουλευτικών εκλογών. Και γι' αυτό λοιπόν τα πολιτικά κόμματα είπαν με απόλυτη σαφήνεια ότι εντάξει ε, θα σας βοηθήσουμε να φτιάξετε μια καινούργια πόλη. Και γι' αυτό το λόγο είχαμε και τη στεναρή υποστήριξη της ε, εθνικής κυβέρνησης. Η κυβέρνηση δεν ήθελε να κάνει λάθος. Ε, ήθελε να έχει μια καλή πολιτιστική πρωτεύουσα και γι' αυτό το λόγο ε, ξεκίνησε σε εμά αυτή η συζήτηση ε, κατά πόσον θα βαδίζουμε εκ του ασφαλούς ή κατά πόσον θα πειραματιστούμε. Αυτό εξηγεί και τον ε, μεγάλο αριθμό των επισκεπτών που είχαμε. Για μας ο πειραματισμός βέβαια είναι πιο σημαντικός. Κατά τα άλλα στο ΠΕΤΣ είχαμε και πάρα πολλές αλλαγές στην στο επίπεδο του management, αλλά εν συνέχεια manager. Ε, κατά τη φάση εφαρμογή ε, ε, πρέπει να σα πω, άλλαξε και ο Δήμαρχο και τα πράγματα δεν ήταν και τόσο εύκολα. Τώρα, κατά πόσον η πόλη είναι ορατή, κοιτάξτε, το Πίτς είναι περίπου 30 χιλιόμετρα από την Κροατία. Κροατία, Σερβία, Σλοβενία. Με αυτές τις χώρες έχουμε ουσιαστική πολιτιστική ανταλλαγή και με τους Γερμανούς λόγω της ε, γερμανικής μειονότητας. Αλλά ε, υπάρχει σαφώς η πολιτιστική διάσταση στη δική μας την πόλη. Τώρα πλέον η πόλη μας είναι πολύ πιο διεθνής από ό,τι ήταν ε, κατά το παρελθόν. Τώρα, τα πέντε χρόνια της ε, προετοιμασίας. Κοιτάξτε, νομίζω ότι οι πόλεις στην ε, φάση της ε, προετοιμασίας θα πρέπει να είναι προοδευτικές, να πειραματίζονται. Γι' αυτό είναι καλό να έχουν αυτά τα πέντε χρόνια της προετοιμασίας. Βεβαίως, πρώτα απ' όλα, θα πρέπει να υπάρχει ένα σταθερό management από το ε, αργή και μετά πρέπει να λάβει κανείς σοβαρά υπόψη του το capacity building και για την ομάδα και για την πόλη να αποκτηθούν ε, ικανότητες ε, και κατά αυτήν την περίοδο θα πρέπει να υπάρχει και το θάρρος της αποτυχίας. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή ίσως θα είναι μια καλή απόφαση. Έτσι τη χαρακτήριζα. Πρόεδρος, πολύ ωραία. Ε, τώρα, ε, στο δεύτερο γύρο ερωτήσεων που θέλετε να υποβάλλετε, θα ήθελα να σας δώσω τη δυνατότητα να ερωτήσετε και μετά να κλείσουν όμως οι ερωτήσεις. Γιατί έχουμε άλλους δύο εμπειρογνώμονες που θέλουν να λάβουν το λόγο και αν έχετε ερωτήσεις και άλλες ερωτήσεις θα μπορείτε να τις κάνετε εκ των υστέρων. Γιατί αν δεν το οργανώσουμε έτσι ε, θα το χάσουμε το παιχνίδι. Πολύ ενδιαφέρουσα όλη η συζήτηση αλλά κάπως πρέπει να παραμείνουμε και οργανωμένοι γιατί έχουμε και χρονικούς ε, περιορισμούς. Ματίτς, Μπιλβάο, Χάιντε και Μπότσκο.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 Ε, είπατε και κάτι το οποίο εγώ ήθελα να ρωτήσω και ε, απαντήστε μου αν έχετε χρόνο πώς ε, εξασφαλίζεται την βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την ε, πολιτιστική πρωτεύουσα. Επίσης, είναι δυνατόν να ε, συνεχιστεί η υλοποίηση τέτοιων δραστηριοτήτων μετά το πέρας της πολιτιστικής πρωτεύουσας. Ποιος είναι ο ενδεχόμενος κίνδυνος της υλοποίησης τέτοιων προγραμμάτων για τις πολιτιστικές πρωτεύουσες, εσωτερικός ή εξωτερικός. Μπορείτε να μας περιγράψετε λίγο τα στοιχεία αυτά. Ε, σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μπιλμπάου. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολλές ερωτήσεις υποβλήθηκαν στον πρώτο γύρο και εγώ ε, το λίγο χρόνο που έχω στη διάθεσή μου θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους υπεύθυνους των πολιτιστικών πρωτευουσών για τη δουλειά που έχουν κάνει. Θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τον Χαβιέρ ε, γιατί ε, κατάφερε να μεταφέρει στη Δονόστια ακριβώς αυτό τον ενθουσιασμό που είδαμε και εδώ. Και πραγματικά ήταν η περηφάνεια της πόλης. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πέρα από αυτό όμως θα ήθελα να ρωτήσω αυτή η ευαισθησία ε, για την Ευρώπη ε, παρέμεινε, αλλά ε, μεταβλήθηκε με οποιοδήποτε τρόπο η πόλη. Δηλαδή, οι, οι, κάτοικοι, οι πολίτες βλέπουν κάποια τροποποίηση, κάποια αλλαγή μετά από την πολιτιστική πρωτεύουσα τι έμεινε για τους κατοίκους, τι άλλαξε για τους ε, κατοίκους. Τώρα κοιτάξτε, εγώ δεν ε, είμαι από την Δονόστια, αλλά είμαι Βάσκα. Ε, και πραγματικά πρέπει να πω ότι αυτή η αυτή την αλλαγή την έζησαν όλοι οι πολίτες γιατί κατάφεραν να περάσουν στους πολίτες, να, να, τους, ε, να τους εμπλέξουν ε, σε μια σειρά από δραστηριότητες ε, και πραγματικά ελπίζω κάτι ανάλογο να ζήσουν και οι άλλες πόλεις. Και επίσης στην, στο Intergroup Μειονοτήτων ακούσαμε αυτό το πρόγραμμα και πέρα από ε, το, τη λευκή βίβλο που ενδεχομένως θα μπορούσε να υπάρξει, κάτι πιο απλό, που θα μπορούσε ίσως να ε, δίνει η μία πόλη στην άλλη. Γιατί βεβαίως ε, το δίκτυο είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά υπάρχει και κάτι άλλο έτσι ώστε να προχωρήσει αυτή η ιδέα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ομιλητές ε, γιατί μας έδειξαν ότι οι πολιτιστικές πρωτεύουσε στην ουσία ε, κάνουν, προωθούν κατά κάποιο τρόπο την Ευρώπη ε, και βελτιώνεται η εικόνα της Ευρώπης στους πολίτες. Είδαμε έκπληξη τους, το, το προπολογισμό στο Πίλσεν όπου από 4,9 εκατομμύρια που θα έπρεπε να είναι ο προϋπολογισμός τελικά ε, ε δόθηκαν πολύ λιγότερα. Ε, μας είπατε ότι 48,6 εκατομμύρια δώσατε για, την, για τις υποδομές. Εκεί υπήρχε ποσοστό συμβολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, τι είδους ήταν και από ποιο ταμείο βγήκαν τα χρήματα. Η κυρία Ποσκόρ. θα μιλήσω ουγγρικά. Ευχαριστώ λοιπόν όλους στο πάνελ για τις ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις. Δύο ερωτήσεις έχω. Πρώτον, είναι πρώτη φορά που άκουσα για αυτήν την άτυπη ομάδα όπου ανταλλάσσονται εμπειρίες και πληροφορίες. Ρωτάω λοιπόν, μήπως θα μπορούσε να τυποποιηθεί αυτή η σχέση Δηλαδή βάσει της εμπειρίας σας, ίσως θα μπορούσατε να υποβάλλετε προτάσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να γίνει το πρόγραμμα αυτό πιο αποτελεσματικό ακόμα. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Η δεύτερη. Το πρόγραμμα όσον αφορά το περιεχόμενό του είναι πια σταθερό και στέρεο. Οπότε, όταν αυτό γίνεται την πρώτη χρονιά και έχουν περάσει μετά πέντε χρόνια και είμαστε στην πέμπτη χρονιά, τι αλλαγές υπάρχουν, ε, υπάρχει περίπτωση να αλλάξει δηλαδή το πρόγραμμα επειδή έχουν περάσει τόσα πολλά χρόνια. Ωραία, προτείνω, όπως κάναμε και πριν, να ακούσουμε τις απαντήσεις. Παρακαλώ. Ε, με την ανάποδη σειρά. Καλά. Ωραία. Εντάξει, εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Σύντομα θα απαντήσω. Η βιωσιμότητα των προγραμμάτων είναι και το μυστικό, κατά τη γνώμη μου. Να συνδέονται δηλαδή με παράγοντες οι οποίοι παραμένουν στην πόλη. Αν όλη τη δουλειά την κάνει η πολιτιστική πρωτεύουσα, τότε έρχεται κάποιος και μετά φεύγει. Δεν είναι καλό αυτό. Πάνω από το 5% των προγραμμάτων που αποτέλεσαν μέρος στο περιεχόμενο του Σεμπαστιάν 2016 παραμένει. Εξαφανίστηκαν ε, προγράμματα που είχαν να κάνουν με την πολιτιστική πρωτεύουσα. Αλλά το κύριο μυστικό για να λειτουργήσει το θέμα είναι να υπάρχουν πιο μόνιμοι αντιπρόσωποι. Και ευχαριστώ πάρα πολύ την ε, Ευρωβουλευτή από τη χώρα των Βάσκων. Πράγματι, και ευχαριστώ πολύ και για τα καλά σας ε, λόγια. Τώρα απαντώ συγχρόνω και στην κυρία Μποσκόρ. Ναι, υπήρξε προσπάθεια να δημιουργηθεί το δίκτυο, αλλά δεν τα καταφέραμε. Ζητήσαμε και βοήθεια. Δεν πέτυχε όμω η προσπάθεια. Και θέλω να σα το πω ότι ορισμένοι θεωρούμε ότι είναι σημαντικό, ίσω, όχι όλοι. Υπάρχουν απόψεις που λένε ότι θα πρέπει να είναι πιο ελεύθερο, πιο χαλαρό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση πάντως έγιναν προσπάθειες να γίνει και κάποια πιο σε βάθος ανάλυση όσον αφορά τις πολιτιστικές πρωτεύουσε. Κατά τη γνώμη μου πάντως, είμαστε το πιο ε, παλιό ε, πρόγραμμα πολιτιστικό στην Ευρώπη. Τώρα για τη χρηματοδότηση που πήραμε στο Σαν Σεμπαστιάν, ήταν μια περίεργη, ιδιαίτερη περίπτωση, γιατί εμεί δεν ζητήσαμε βοήθεια για υποδομέ. Το πρόγραμμά μα βασιζόταν στη συνύπαρξη. Και το Σαν Σεμπαστιάν είναι μια πόλη που τουριστικά μιλώντα ποτέ δεν είχε παρουσιαστεί αλλιώ. Δεν το έκανε για να τραβήξει τουρισμό. Έχει. Το 90% απασχολείται στον τουρισμό το καλοκαίρι. Άρα δεν πρόκειται για την ίδια περίπτωση. Εμεί θέλαμε να έρθει ο να γνωρίσει, να καταλάβει την Ευρώπη. Και πετύχαμε για πρώτη φορά να έχουμε δύο βοήθειες από τη Δημιουργική Ευρώπη και η μία τέλειωσε πολύ πρόσφατα. Αυτά είχα να πω. Ε, ο κύριος Σούτσανεκ. Speaking about the, the financing and... Σχετικά με την χρηματοδότηση και την βιωσιμότητα. Κατά τη δική μου άποψη, ε, ο καλύτερος τρόπος είναι ε, η οικοδόμηση ικανοτήτων, capacity building, δηλαδή να η κοινή δουλειά ε, στη διάρκεια της προετοιμασίας του διαγωνισμού και μετά την επιτυχία στον διαγωνισμό ε, κατά την άποψή μου αυτός είναι ο τρόπος ε, να επιτύχει κανείς αλλά και να διατηρήσει βιώσιμη χρηματοδότηση. Και πιστεύω ότι θα πρέπει κανείς ε, να αναζητά μελλοντικές πηγές χρηματοδότησης ε, από πόλεις οι οποίες ολοκληρώνουν την ε, δράση τους ε, και ενδεχομένως και μια ανοιχτή πρόσκληση για το 2020 ε, να ε, χρησιμοποιηθούν τα χρήματα για τις legacy activities, ε, συγκεκριμένοι τρόποι έτσι ώστε να παραμείνει το κληροδότημα και μετά την πάροδο της προλητιστικής πρωτεύουσας. Το πρόβλημα που ανέφερα εγώ προηγουμένως είναι οι προσδοκίες που έχουν οι πολίτες να δείξουν την διαφορετικότητα της ε, πόλης τους ε, και από την άλλη μεριά το γεγονός ότι πολύ συχνά τα προγράμματα ε, βασίζεται σε μια εθνική ή διεθνή ή ευρωπαϊκή βάση, επί τη βάση δηλαδή διεθνών ή ευρωπαϊκών αρχών. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει μια αίσθηση έλλειψης ισορροπίας. Πάντως, ε, σίγουρα θα έχετε και τη δυνατότητα να αλλάξετε ορισμένα πράγματα στη φάση υλοποίησης. Εκεί μπορείτε να ξεκινήσετε με ανοιχτούς διαγωνισμούς ε, για σύγχρονο design, πάντα όμως ε, επί τη βάση των αναγκών των απλών καθημερινών πολιτών της πόλης. Κοιτάξτε, πέντε χρόνια είναι ένα μεγάλο διάστημα για την ανάπτυξη των projects και θα έλεγα και εγώ ότι θα πρέπει λίγο να ε, είναι πιο βραχία η περίοδος. Πάντως έχετε ένα μπούσουλα, στο πούμε, έχετε ένα, μια σύμβαση και αυτή την σύμβαση θα πρέπει να την ακολουθήσετε ε, ε, με συχνή επιτήρηση έτσι ώστε να μην εκτροχιαστεί η πόλη πώς αλλάζει η πόλη, πώς άλλαξε η πόλη στην περίπτωση του Πίλσεν. Άλλαξε με συγκλονιστικό τρόπο. Οι άνθρωποι, ας πούμε, άρχισαν ε, στο Πίλσεν να χρησιμοποιούν το δημόσιο χώρο. Ε, σε πολλές χώρες ε, είναι φυσικό να ζει κανείς έξω, να ζει στους δρόμους, στις πλατείες. Στην περίπτωση του Πίλσεν όμως, η πιο ορατή αλλαγή ήταν ότι ε, ο πολιτισμός, η κουλτούρα βγήκε από τους κλειστούς τείχους των κτηρίων και βγήκε στους δρόμους. Οι άνθρωποι απέκτησαν περιέργεια για το τι συμβαίνει γύρω τους. Και η συμμετοχή επίσης, ε, ο βαθμός συμμετοχής, κάτι απολύτως καινούριο, με μεγάλο αντίκτυπο στην πόλη. Τελευταίο, όσον αφορά τις υποδομές, 48 εκατομμύρια για ε, την υποδομή μιας πόλης 170.000 κατοίκων ε, είναι πολύ. Λιγότερο από 20% ε, ήταν η συμβολή των διαφορετικών ταμείων. Και δεν ξέρω αν το μήνυμα αυτό είναι καλό ή κακό, αλλά όσον αφορά την πολιτική συνοχής, η τσεχική την πολιτικη συνοχή, η άρχισε να θεωρείται αναπτυγμένη χώρα, επομένως δίνονται λιγότερα χρήματα για την πολιτιστική ε, παραγωγή. Δεν είναι το ίδιο όμως για την Κροατία. Η εντύπωσή μου πάντως είναι ότι η Ριέκα τα πάει πάρα πολύ καλά όσον αφορά το ισοζύγιο, αυτή την ισορροπία ανάμεσα σε projects που αφορούν τις υποδομές και τα άλλα που δεν αφορούν υποδομές τα οποία ονομάζουμε συνήθως soft projects. Επίσης, ε, διαπίστωσα ότι δημιουργούνται κάποιες νέες γειτονιές, δημιουργικές γειτονιές και πιστεύω ότι αυτό εν τέλει ε, θα αποδειχθεί ελπιδοφόρο και ε, επιτυχές. Νομίζω πραγματικά ότι η ΡΕΚΑ είναι σε πολύ καλή τροχιά, σε πολύ καλό δρόμο. Ευχαριστώ πολύ. Βρισκόμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο και όσον αφορά τη βιωσιμότητα ε, είμαι ε, πεπισμένος ότι υπάρχουν και καλά και λιγότερα ε, καλά παραδείγματα. Τη βιωσιμότητα την επιτυγχάνει κανείς δημιουργώντας βιώσιμες υποδομές και επενδύοντας σε ανθρώπους. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ε, στο ΠΕΤΣ μπορούσαμε να φτιάξουμε υποδομές, ε, όχι μόνο αυτές που προανέφερα, αλλά κατ' ουσίαν στο ΠΕΤΣ μετά το 2010 δεν διαλύθηκε το management. Γιατί μέσα στο management είχαμε και όλα τα έργα υποδομής. Δηλαδή τα έργα υποδομής δεν είχαν ε, τοποθετηθεί στο ε, Δημαρχείο, αλλά σε εμά στο management. Και αφού ε, τέλειωσε η πολιτιστική πρωτεύουσα, αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε περαιτέρω αυτή την εμπειρία που είχαμε συγκεντρώσει και το πολιτιστικό τμήμα του management ε, μετά μετατράπηκε η εταιρεία που λέγεται Εταιρεία Ανάπτυξης της Πόλης. Και υπάρχει και μέχρι σήμερα. Αυτοί είχαν συγκεντρώσει ε, πολύ καλή εμπειρία, κυρίως όσον αφορά την ε, απόκτηση ενωσιακών κονδυλίων. Κατά τα άλλα, όσον αφορά το καλλιτεχνικό κομμάτι, το παλιό management ε, αφομοίωσε όλα τα παλιά Ινστιτούτα, τα πολιτιστικά, αν ήταν καλό ή όχι. Τώρα δεν μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό. Αλλά, με πάση περιπτώσει, με αυτόν τον τρόπο η πόλη μπόρεσε να επιτύχει ε, βιωσιμότητα των υποδομών και νομίζω ότι τελικά αυτό είναι καλό. Όσον αφορά τη φάση εφαρμογή, ακούσαμε πάρα πολλά. Εγώ το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να υπογραμμίσω ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια καλή ισορροπία ανάμεσα σε τοπικούς φορείς οι οποίοι ενδεχομένως δεν είναι τόσο ορατοί ή δεν εφαρμόζουν μεγάλα προγράμματα ισορροπία ανάμεσα στους τοπικούς και τα μεγάλα εξωτερικά ονόματα. Ε, αυτό ε, πρέπει κανείς να το μελετήσει βέβαια πολύ προσεκτικά να υπάρχει όπως σας είπα αυτή η ισορροπία. Και ένα άλλο στοιχείο που θέλω να αναφέρω σχετικά με τη φάση της ε, εφαρμογής. Από την δική μου εμπειρία μπορώ να σας πω ότι αν δεν είναι καλά οργανωμένη η επικοινωνία με τους πολίτες, τότε τα πράγματα ε, μπορούν να εξελιχθούν πολύ αρνητικά. Ε, θα πρέπει κανείς να εξηγήσει στους πολίτες τι κάνει, πώς το κάνει, ποιοι είναι οι κίνδυνοι. Αυτή λοιπόν η επικοινωνία με τους πολίτες είναι καθοριστική σημασία για τις επενδύσεις 140 εκατομμύρια επενδύθηκαν και το 85% ήταν ε, χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολύ μεγάλο δηλαδή το ποσοστό. Ε, και τέλος, αυτό που πρότεινε η κυρία Πότσκο. κοιτάξτε, εγώ είχα την ε, τιμή να συνειδρύσω αυτό το άτυπο δίκτυο. Το υπενήχθηκα αυτό προηγουμένως. Ε, σας το είπα ότι τότε υπήρχε αυτή η ανάγκη να συζητάμε μεταξύ μας το τι είναι μια πολιτιστική πρωτεύουσα και πώς μπορεί κανείς να την επιτύχει με επιτυχία. Και φτιάξαμε μια πολιτική, τώρα πια είμαστε μια ε, εταιρεία, ε, είμαστε ε, κλειστοί πλέον, παραμένουμε μεταξύ μας, αλλά τα πρώτα χρόνια είχαν ε, συμπεριληφθεί ε, δύο-τρεις πολιτιστικές πρωτεύουσες σε αυτό το δίκτυο και τότε ετίθεται ακριβώς σε αυτό το θέμα. Γιατί υπάρχουμε, για ποιο λόγο. Αυτή είναι μια διαδικασία, ένα επίκαιρο ερώτημα, αλλά όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, εφόσον ληφθεί η απόφαση να ε, θεσμοθετηθούμε, τότε νομίζω ότι ε, πρέπει κανείς ε, να δεχτεί αυτή την άποψη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ως εκ τούτου κλείσαμε το πρώτο γύρο των παρεμβάσεων και θα περάσουμε τώρα στο δεύτερο. Και θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Διάνα Σίβιλε. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω λετωνικά. Ευχαριστώ λοιπόν. Η Ρήγα ήταν το 2014 Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα. Και ήταν πάντα στο σταυροδρόμι ανάμεσα το βορρά και τον νότο, την Ανατολή και τη Δύση. Πάντα δημιουργούσαμε επίσης δρόμους. Κάποια στιγμή είχαμε φτιάξει του και χρυμπαριού το δρόμο, που ήταν ο εμπορικός δρόμος που περνούσε από την Ρήγα. Και ακριβώς και χρυμπάρι εμπορευόμασταν, που είχε πολύ μεγάλη προστεθέμενη αξία εκείνη την εποχή. Η Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα λοιπόν πρέπει να δημιουργεί δρόμους και τρόπους. Και εμείς ακριβώς αυτό ε, προσπαθούμε να δούμε πώς να περάσει το σημερινό μήνυμα και σκεφτήκαμε πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό. Το δικό μας πρόγραμμα δημιουργήθηκε ήδη από την οικονομική κρίση που ήταν μια έκτακτη περίοδος ε, για μας γιατί ολόκληρη κοινωνία βρισκόταν σε κατάθλιψη και η κοινωνία χρειαζόταν ε, κάτι κάπου για να πιαστεί. Και γι' αυτό και εμείς προσφέραμε το πρόγραμμα αυτό, Force Majeure, κατάσταση έκτακτης ανάγκης και πήγε καλά. Γιατί θεωρήσαμε ότι ο πολιτισμός είναι αυτό ακριβώς από το οποίο μπορεί κανείς να πιαστεί, που μπορεί να βοηθήσει όλους να αλλάξει την πόλη, να κάνει τον κόσμο να γνωριστεί ο ένας με τον άλλον κτλ. Έτσι λοιπόν, πιστεύω ότι πολλά έχουμε να κερδίσουμε από την εμπειρία αυτή. Από τη βασιστήκαμε σε, κάποιους, ε, σε κάποια θέματα, σε κάποιους τίτλους που μας επιτρέπουν έτσι να διαμορφώσουμε καλύτερα το πρόγραμμα. Πρώτα απ' όλα, ο πρώτος πυλώνας για μας ήταν ο ωκεανός. Στο θεματικό αυτό σκέλος συζητούσαμε για τις ανθρώπινες αξίες, για την κατανόηση. Υπήρχαν ε, δραστηριότητες και συμμετοχή σε διάφορα κοινωνικά επίσης προγράμματα. Ένα άλλο ε, μεγάλο παιχνίδι που είχαμε κάνει ήταν ε, συζητήσεις που είχαμε για την ε, κοινή κουλτούρα της Ευρώπης, για θέματα ελευθερίας, εξουσίας. Κοιτάξαμε τι είχε γίνει τα προηγούμενα χρόνια ε, με τους πολέμους και πώς άλλαξε η Ευρώπη μετά τον πόλεμο, το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Freedom Street, το λέγαμε. Πολύ σημαντικό για τη Ρίγα αυτό. Το τρίτο θέμα ήταν roadmap. Ήταν ο χάρτης πορείας. είδαμε τι μεγάλο κέρδος είχαμε από την πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Η κοινωνία όντως είχε αλλάξει, έγινε περισσότερο ανοιχτή και ο κόσμος ασχολήθηκε πολύ περισσότερο με τον πολιτισμό. Όταν ξεκινήσαμε είδαμε τις στατιστικές και καταλάβαμε ότι μόνο 15% του κόσμου συμμετέχει. Και γι' αυτό αποφασίσαμε να έχουμε επικοινωνία για την πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης και ακριβώς να απευθύνεται στο υπόλοιπο 85% που ουσιαστικά αποτελούν και αυτοί δυνητικά καταναλωτές πολιτισμού. Έτσι λοιπόν, συμμετείχε η πόλη σε αυτή την προσπάθεια, κάτι που βοήθησε ο κόσμος να συνειδητοποιήσει περισσότερο περί τίνος πρόκειται. Ακολούθησαν κι άλλες αποφάσεις από το Δήμο. Αλλάξαμε την πολιτιστική στρατηγική της Ρήγα. Δουλέψαμε με διάφορες κοινότητες στα προάστια αλλά και στο κέντρο. Και είναι μια δουλειά που συνεχίζεται ακόμα και σήμερα γιατί ήταν πολύ καρποφόρα. Έχουμε δημιουργήσει στην πόλη διάφορα πολιτιστικά κέντρα και το πιο σημαντικό έγινε, δηλαδή ότι αυξήθηκε η πρόσβαση του κοινού σε πολιτιστικά δρόμενα. Όταν μιλάμε όμως για αυτούς τους δρόμους, τους διάφορους, είπαμε του και πρώτα απ' όλα, όλα αυτά τι συμβολίζουν. Συμβολίζουν οι δρόμοι, συμβολίζουν τις σχέσεις. Ε, είτε με την υπόλοιπη Ευρώπη, είτε στην περιοχή. Όπως είπαμε, αναπτύχθηκε περισσότερο η πολιτιστική δραστηριότητα και δημιουργήθηκε ένα δίκτυο όχι μόνο με εκπροσώπους του πολιτισμού, αλλά και με κόσμο από άλλους τομείς. Δημιουργήθηκαν συνέργειες δηλαδή. Και κάτι άλλο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εμείς γιορτάζουμε τον πολιτισμό, γιορτάζουμε την ποικιλομορφία στον πολιτισμό επίσης. Κάτι το οποίο προωθεί την κατανόηση μεταξύ των διαφόρων κοινότητων στη χώρα. Οι στατιστικές πάντως είναι πάρα πολύ θετικές. Εδώ βλέπετε τα νούμερα που μιλάνε από μόνα τους. Το πρόγραμμα ήταν ιδιαίτερα επιτυχές. Αυξήθηκαν οι τουρίστες, οι επισκέπτες, έγινε περισσότερο γνωστή η πόλη της Ρήγας στο εξωτερικό ήρθαν διάφορα τηλεοπτικά συνεργεία και γύρισαν σκηνές που μετέδωσαν στη συνέχεια στις χώρες τους. Ναι, αυτή είναι η οικονομική πτυχή, συμφωνώ, που εύκολα μπορεί κανείς να την εκφράσει ποσοτικά. Αλλά θα ήθελα να αναφέρω και ένα ακόμα παράδειγμα που έχει να κάνει με την οικονομική πτυχή που δεν γίνεται πάντα κατανοητό ή δεν το καταλαβαίνει αρκετά ο κόσμος. Στη Ρήγα, και εδώ θα σας δείξω μια άλλη εικόνα, εδώ είχαμε ένα διαγωνισμό ε, τραγουδιού. 20.000 τραγουδιστές από πάρα πολλές χώρες συμμετείχαν. Και εδώ βλέπετε τη σκηνή που βρίσκεται, ε, είναι ανοιχτή. Και βλέπετε όλους τους τραγουδιστές εδώ. Ήτανε υπό την αιγίδα της UNESCO. Και τώρα όμως είχαμε από 73 χώρες τραγουδιστές που ήρθαν και τραγούδισαν στο φεστιβάλ μας. Κοιτούμε φυσικά και τις οικονομικές συνέπειες τέτοιων εκδηλώσεων και καταλάβαμε ότι 3 εκατομμύρια είχαμε επενδύσει, τα οποία είχαν μεγάλη η οικονομική επίπτωση, αλλά κερδίσαμε 21,5 εκατομμύρια. Να λοιπόν ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα του πολιτισμού, ο οποίος είναι πολύ πιο ισχυρός από ό,τι μπορεί κανείς να φανταστεί εκ πρώτης όψεως. Πάντως, ναι, πάντα πρέπει να σκεφτόμαστε την οικονομική πτυχή. Συγχρόνως όμως, το συναισθηματικό κέρδος είναι επίσης πολύ μεγάλο από τέτοιου είδους εκδηλώσεις πολιτιστικές. Και γι' αυτό σας δείχνω και την επόμενη εικόνα που την δείχναμε στην αρχή και αποτελεί μία λυσίδα. Τον Ιανουάριο το κυκλοφορήσαμε αυτό. Ήταν μια ζωντανή αλυσίδα ε, ανθρώπων που διαβάζουν βιβλία, που αγαπάνε τα βιβλία. Για τέσσερις ώρες λοιπόν ήμασταν στους δρόμους και μεταφέραμε βιβλία από το παλιό κτίριο της βιβλιοθήκης στην νέα βιβλιοθήκη, το νέο κτίριο που το βλέπετε εδώ και ονομάζεται ε, ο πύργος της ζωής. Αυτή η ανθρώπινη λυσίδα λοιπόν ήταν κάτι συναισθηματικά πάρα πολύ φορτισμένο, γιατί ήταν ένα σωρό κόσμο στο δρόμο που περνούσαν τα βιβλία από χέρι σε χέρι για να μεταφερθούν από το παλιό κτίριο στο καινούριο πολύ δυνατή στιγμή και τέτοιες στιγμές έχουν μεγάλη σημασία και από αυτές κερδίζει κανείς ακόμα περισσότερα. Τώρα πέντε χρόνια μετά ε, προσπαθώ να απαντήσω κι εγώ στον εαυτό μου ε, στην ερώτηση τι είναι το τόσο μοναδικό με τις ευρωπαϊκές ε, πολιτιστικές πρωτεύουσες. Οπότε πρώτα απ' όλα είναι η προοπτική που περιμένει στην πρωτοβουλία αυτή να υλοποιηθεί. Αυτό είναι ήδη ένα μεγάλο κέρδος. Και είναι πολύ σημαντικό επίσης στα πλαίσια ε, αυτού του εθνικού περιβάλλοντος ε, που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για ένα μοσαϊκό πολιτισμών. Η εκπαίδευση, οι επιστήμες βέβαια έτσι καλλιώς έχουν ε, κυρίαρχο ρόλο στις διάφορες ανταλλαγές, αλλά υπάρχουν και όλες οι άλλες αξίες που γνωρίζουμε. Πάντως για μας, και αυτό ακριβώς συμβολίζει και το πρόγραμμά μας που το ονομάσαμε έκτακτη ανάγκη, είναι ότι έχουμε κάποιες αξίες, κάποιους αλγορίθμους και όλες τις πολιτιστικές μας αξίες τις βάζουμε σε ένα τέτοιο πρόγραμμα. Συγχρόνως όμως υπάρχει και μια κοινωνική εμπειρία στο θεσμό αυτό πολιτιστικής πρωτεύουσας. Γιατί ο πολιτισμός τότε συνδέεται και με άλλες πτυχές και με άλλες αξίες. Στη δικιά μας την περίπτωση λοιπόν δείξαμε ότι ο πολιτισμός είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο για την Λετωνία, αλλά και ο λετωνικός πολιτισμός για ολόκληρη την Ευρώπη. Γιατί όλοι όσοι συμμετείχαν σε ένα τέτοιο πρόγραμμα, είτε σαν παράγοντες είτε σαν θεατές, αναγνώρισαν την αξία του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τελευταία στο πρώτο ε, μπλοκ κυρία Ροσέλα Ταραντίνο, η οποία μας παρουσίασε την πολιτιστική πρωτεύουσα ματέρα και χαίρομαι πάρα πολύ που σας δίνω το λόγο. Yes, Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση που μου απευθύνατε. I'm speaking about the current θα μιλήσω για την ε, Ματέρα που είναι η φετινή πρωτεύουσα, πολιτιστική πρωτεύουσα. Η Ματέρα είναι μια πόλη ε, που έχει υποστεί πάρα πολλές ε, αλλαγές και τροποποιήσεις. Φαίνεται ότι πιστεύετε ότι είχε το σχήμα της Ιταλίας ε, και βεβαίως ε, έχει γίνει και ε, πολιτιστική κληρονομιά στα πλαίσια της UNESCO. Εξαιρετικές προσωπικότητες από την διεθνή σκηνή αλλά και σε τοπικό επίπεδο έχουν επισκεφθεί τη ματέρα. Βεβαίως ο διαγωνισμός όμως για τον τίτλο ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό γιατί αυτός ο διαγωνισμός έδωσε τη δυνατότητα ή μάλλον όθησε τους ε, ντόπιου ε, να οικοδομήσουν ένα συλλογικό κλίμα. Δεν ήταν ένα όνειρο απλώς ή δεν ήταν απλώς μια συγγραφή υποχρεώσεων όσο εξαιρετικό και αν θα ήταν ε, αυτό, αυτή η δέσμη, ας πούμε, το τεύχος συγγραφή συγγραφής ε, ε, υποχρεώσεων, αλλά ήταν ε, μια ιδέα για την πόλη σου με ταυτόχρονη υποβολή ερωτημάτων που δεν ήταν πάντα εύκολα σε συνεργασία και με άλλους καλλιτέχνες από όλη την Ευρώπη. Εμείς πραγματικά τότε καταλάβαμε ότι ξεκινούσε μια πολύ μεγάλη ε, αλλαγή. Όταν ε, πήραμε στα χέρια μας ε, τα τεύχη της εγγραφής υποχρεώσεων, πραγματικά καταλάβαμε τι συμβαίνει. Η Ματέρα είναι μια μικρή σχετικά πόλη με 60.000 κατοίκους. Είναι μια τυπική μικρή πόλη της Ευρώπης σε μια περιφέρεια η οποία δεν, έχει πυκνή, δεν είναι πυκνοκατοικημένη όπως συμβαίνει και σε άλλες περιφέρειες της Ευρώπης. Μπορεί ε, μια πόλη η οποία μέχρι τώρα δεν είχε δημιουργήσει πολιτισμό αλλά ε, κατανάλωνε πολιτισμό που είχε δημιουργηθεί αλλού να δημιουργήσει δικό της. Ναι, η απάντηση είναι θετική και μπορεί να δημιουργήσει και ένα νέο ακροατήριο. Και ε, εμείς λοιπόν αποφασίσαμε ότι πολύ σοβαρά θα παίρναμε υπόψη ε, αυτό το πολιτιστικό έτος ή θα έλεγα καλύτερα αυτά τα έτη της προετοιμασίας. Ε, επομένως κάναμε και εισαγωγή πολιτιστικών ε, αγαθών αλλά και κάναμε και παραγωγή. Ε, επίσης αποφασίσαμε όχι μόνο να κάνουμε δική μας στη ματέρα παραγωγή πολιτιστικών προϊόντων, αλλά και να δημιουργήσουμε και προϋποθέσεις για μελλοντική παραγωγή. Γι' αυτό ξεκινήσαμε, ιδρύσαμε το Open Design School της Ματέρα, που ε, δημιουργεί το setup ε, για πολλές εκδηλώσεις, για πολλές εκθέσεις, ε, έτσι ώστε ο δημόσιος χώρος να εννοηθεί με διαφορετικό τρόπο. Η ματέρα δεν ήταν απλώς μια σκηνή, αλλά αποτέλεσε ένα εργαστήριο παραγωγής που χρησιμοποίησε την τοπική σκηνή, τους τοπικούς καλλιτέχνες, αλλά και πολλούς ε, διεθνούς ε, φήμης ε, καλλιτέχνες. Και βέβαια πάνω απ' όλα 70% της εργασίας έγινε σε συνεργασία με τους πολίτες οι οποίοι έδειξαν να συμμετέχουν με μεγάλο ενθουσιασμό. Έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα. Ας πούμε, έχουμε την λυρική όπερα ε, που είδαμε και στο Άρτε. Στην ουσία όμως είχαμε παραστάσεις όπερας εκτός της λυρικής σκηνής αλλά εντός της πόλεως με συμμετοχή όλων των πολιτών. Ε, είχαμε το πρόγραμμα Social Lights όπου οι πολίτες αποφάσισαν να δημιουργήσουν ε, φώτα και να τα δείξουν στην ε, εναρκτήρια τελετή και πήγαμε μάλιστα και σε ε, άλλα μέρη όπως είναι νοσοκομεία, σχολεία, ε, σχολεία χορού κλπ. Έτσι ώστε όλοι να παίξουν, να συμβάλλουν σε αυτό το παιχνίδι της πολιτιστικής παραγωγής. Εδώ έχουμε ένα άλλο παράδειγμα οι άνθρωποι έδειξαν τις συλλογέ τους, ε, οτιδήποτε ε, συνέλεγαν ή ήταν αιμονικό για αυτούς. Και ο Βιτζίλιο Σέρνη, ο χορογράφος, ε, τα ένωσε όλα αυτά. Επίσης, πρέπει να πω ότι 400.000 άνθρωποι δημιούργησαν ε, πολίτες, δημιούργησαν την ε, αόρατη πόλη, ε, την πόλη των αισθήσεων, των συγκινήσεών τους και των συναισθημάτων τους. Πολλά, πολλά ήταν τα projects, αλλά υπάρχει κάτι το οποίο με εντυπωσίασε την προηγούμενη Κυριακή. Δουλεύουμε και με τις πιο απομακρυσμένες ε, περιοχές. Ε, ε, έχουμε ένα πρόγραμμα που λέγεται Garden Top και ένας νέος γεωργός από ένα πολύ μικρό χωριό της Μπαζιλικάτα είπε στον καλλιτέχνη δώστε μας τη δυνατότητα να δούμε νέες δυνατότητες που δεν βλέπουμε τώρα και δείξτε μας το μέλλον μας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι αυτή είναι και η ουσία μιας ευρωπαϊκής πρωτεύουσας. Εδώ σας δείχνω ένα άλλο project για τον τουρισμό ε, τουρίστες που θεωρούνται ε, πρόσκαιροι πολίτες. Ε, θα πρέπει τώρα βέβαια να δούμε πώς ε, μπορούμε να, γενικά στην Ευρώπη τους τουρίστες να τους θεωρούμε όχι ξένους, αλλά ε, πολίτες για ένα μικρό διάστημα. Ε, ε περίπου 2 εκατομ... δισεκατομμύρια views είχαμε στα προγράμματα της Ματέρα και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, να ε, πούμε ότι πρόκειται για πολύ επιτυχημένη πρωτοβουλία. Ε, αυτό το είπατε και εσείς, το είπαν όλοι οι προηγούμενοι ομιλητές. από την άλλη μεριά είναι πολύ σημαντικό ανάμεσα στην ε, Κομισιόν, στην πόλη και την Εθνική Κυβέρνηση να υπογραφεί μια δεσμευτική σύμβαση, γιατί δεν μπορεί να είναι μόνη της ε, η πόλη. επομένω. θεωρώ πολύ σημαντικό αυτό. Επίσης, θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο την ενδυνάμωση της ε, διασύνδεσης και σε ευρωπαϊκό ε, επίπεδο και σε περιφερειακό, δηλαδή και αυτές οι περιφερειακές ευρωπαϊκές πολιτικές είναι πολύ σημαντικές. Εμείς ε, πιστεύουμε και συμφωνώ απολύτως με προλαλήσαντες ε, ότι θα πρέπει να ενδυναμώσουμε πραγματικά την ομάδα των πολιτιστικών πρωτευουσών. Εμείς δημιουργήσαμε, κάναμε μια ε, ομάδα ε, μπάσκετ και έναν αγώνα μπάσκετ της οικογένειας ε, των πολιτικών πρωτευουσών πολιτιστικών πρωτευουσών, συγγνώμη, αλλά πρέπει να είμαστε ομάδες, όχι μονάχα μια οικογένεια. Ε, βέβαια τα προβλήματα είναι πολλά. Υπάρχει άλλωστε και η δημιουργική γραφειοκρατία. Γραφειοκρατία δηλαδή σε οτιδήποτε σχετίζεται με τη δημιουργία. Η επικοινωνία είναι πολύ σημαντική. Πολλά μπορούμε να κάνουμε μαζί σχετικά με τον βιώσιμο τουρισμό που είναι πολύ ε, καλός στόχος, ε, την διανομή κλπ. Ίσως ε, μετά απαντώντας σε ερωτήσεις σας να μπορέσω να μιλήσω παραπάνω. Ευχαριστώ πολύ λέει η Πρόεδρος. Τώρα να υποβληθούν ερωτήσεις από ποιον επιθυμεί. Julie Ward. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να σας ε, ευχαριστήσω. Ευχαριστώ για τις ε, εισηγήσεις που άκουσα και λυπάμαι πάρα πολύ για αυτές που έχασα. Μ' αρέσει πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ, κυρίως ε, διότι άκουσα την εισήγηση από τη ματέρα στην εναρκτία τελετή έπαιξε και ο γιος μου και μου είχε στείλει ένα βίντεο. Είναι δραματουργός, ασχολείται με μουσική. Δυστυχώς εγώ τότε δεν μπόρεσα να έρθω. Ήμουνα σε ταξίδι, αλλά μου έστειλε ένα βίντεο και εκεί ε, φαίνεται απευθύνεται στο κοινό και σκέφτηκα ότι πω πω, για δες, να και ο γιο μου παίζει και αυτό σε μια πολιτιστική πρωτεύουσα. Ήρθε λοιπόν, επέστρεψε πίσω με πολύ θετική εμπειρία από την πολιτιστική πρωτεύουσα Ματέρα και τώρα το χρόνο που έχω θέλω να το χρησιμοποιήσω για να σας πω ότι υπήρξαν και δύσκολες εμπειρίες. Μία εξ αυτών είναι αυτά που έγιναν στις αρχές του έτους στο Πλόβτιβ Εκεί είχαμε μια κατάσταση όπου οι ντόπιοι ε, πολιτικοί ε, ενίσχυσαν την ομοφοβία. Στην πόλη αυτή υπήρχε μία έκθεση για το, την παρέλαση των ομοφιλοφίλων Pride στα Βαλκάνια και οι πολιτικοί προσπάθησαν να παρέμβουν στην οργάνωση αυτού του προγράμματος. Ε, πήρα πληροφορίες σχετικά με αυτό, γιατί εγώ είμαι σε επαφή με το Plovdiv. Ε, το Φεβρουάριο είχαμε πάει και αποστολή. Το θέμα βέβαια δεν ετέθη καθόλου. Έχω όμως φίλους ε, που συμμετέχουν ευρύτερα στο κίνημα και είχα ξαναπάει και το καλοκαίρι που είχαν αυτή την επίθεση την ομοφοβική, μου έστελναν πληροφορίες, αυτές τις φωτογραφίες, με γκράφιτι, ε, τις ε, απειλές που δεχόντουσαν αυτοί που εργάζονταν για το Ίδρυμα. Ξέρω ότι είσαστε αδελφές πόλης και γι' αυτό το θίγω το θέμα. Επίσης, το θέμα που επελέγει για το Πλόπτικ ήταν νομίζω το σύνθημα «Together», «Μαζί». Ας έρθουμε κοντά, είμαστε μαζί. Αυτό είναι ευρωπαϊκή αξία ε, φοβάμαι όμως ότι η ομοφοβία δεν είναι ευρωπαϊκή αξία. Πάντως θέλω να σας πω ότι εγώ τότε ανησύχησα πάρα πολύ γιατί πιστεύω ότι αυτό δεν είναι καλή διαφήμιση για την Ευρώπη, για μια ευρωπαϊκή πολιτιστική πρωτεύουσα. Το να υπάρχει αυτή η αντιευρωπαϊκή διαδήλωση. Και γι' αυτό ερωτώ, εσείς τι μπορείτε να κάνετε. Αν ε, κάνετε κι εσείς αυτή την εμπειρία, τι θα κάνετε. Γιατί το θέμα έφτασε στις εφημερίδες, στο Guardian, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Νομίζω λοιπόν ότι οι άνθρωποι που εργάζονται στο Ίδρυμα ε, έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά στο να υπερασπιστούν το πρόγραμμά τους και νομίζω ότι οι ντόπιοι πολιτικοί που ε, δεν είναι ομοφοβικοί και αυτοί έκαναν πάρα πολύ καλή δουλειά, αλλά κατ' ουσίαν όλοι καλούμεθα να διαφυλάξουμε τις ε, ευρωπαϊκές αξίες, κυρίως ε, όταν παρισφρέει και το ευρωπαϊκό χρήμα και ο ευρωπαϊκός λογότυπος. Αυτή την εμπειρία έκαναμε το με την πόλη που σας είπα, αλλά ανησυχώ λιγάκι και ε, για θέματα λογοκρισίας, ε, γιατί υπήρξαν τέτοιες ενδείξεις και πρέπει να σας πω μια εταιρεία SH αστερίσκος T SH αστερίσκος T είναι μια εταιρεία ε, που ανέλαβε να κάνει κάποια δουλειά στη Βαλέτα και όταν πήγαν εκεί τους είπανε δεν μπορείτε να δουλέψετε εδώ, δεν μπορείτε εκεί, δεν μπορείτε παραπέρα και όλα αυτά είχαν με τη δολοφονία της δημοσιογράφου και κάθε βράδυ ε, βεβηλώνεται κατά κάποιον τρόπο το άγαλμά και το πρωί οι αρχές ε, το ε, καθαρίζουν και πάλι εκ νέου. Τέλος, προέκυψε και ένα έργο θεατρικό ε, για την εμπειρία τους για θέματα λογοκρισίας. Δεν μπόρεσαν να το ανεβάσουν στη Μάλτα, αλλά θα το ανεβάσουν στο Λονδίνο. Εγώ πιστεύω ότι αν δεν είμαστε προσεκτικοί, ε, δημιουργούνται προβλήματα αν δεν προσέχουμε το πώς ε, χρησιμοποιούνται τα χρήματά μας. Τα θίγω αυτά, ε, διότι πρέπει να τα εξετάσουμε. Πρέπει να τα εξετάζουμε ως πολιτική, αλλά να μην ξεχνάμε και τους καλλιτέχνες. Όλα αυτά δεν είναι καλή εικόνα για μας και δεν είναι καλή εικόνα για αυτό το θαυμάσιο δίκτυο που έχετε δημιουργήσει σχετικά με τις επιτυχημένες πρωτεύουσες της Ευρώπης. Ο κύριος Αντάμοφ, παρακαλώ. Εκτός μικροφώνου, δεν τον ακούμε τον κύριο Δέμοφ. Ευχαριστώ. Άκουσα διάφορα ενδιαφέροντα πράγματα και είμαι πολύ ικανοποιημένος από αυτά που έχω ακούσει. Σας συγχαίρω για όλες τις τόσο καλές πρωτοβουλίες που έχετε αναλάβει μέχρι τώρα. Όμως θα ήθελα να υπογραμμίσω δύο πράγματα. Όσον αφορά την ε, δημοσιότητα και τη διαφήμιση, πολλοί λένε ότι δεν είναι αρκετή. Πράγματι και εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε περισσότερα. Μπορούμε να επενδύσουμε πολύ περισσότερο στην ε, διαφήμιση ώστε να προσελκύονται όλο και περισσότεροι άνθρωποι για να παρακολουθήσουν όλα αυτά τα ωραία πράγματα που συμβαίνουν στις πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης. Και κάτι άλλο, αν και μου έχει απαντηθεί λιγάκι. Τι γίνεται, άπαξ, και τελειώσει ο χρόνος κατά τον οποίο μία πόλη είναι πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Γιατί, από ό,τι φαίνεται, κάθε πόλη έχει τις αρχικές της ιδέες, τις δημιουργικές που θα έπρεπε να υλοποιηθούν, αλλά όχι μόνο σαν ένα πυροτέχνημα που ξαφνικά ανάβει και αμέσως μετασβήνει. Πιστεύω ότι πρέπει να σκεφτούμε, να δημιουργήσουμε μια πλατφόρμα, ένα δίκτυο που να μπορεί να χρησιμεύσει και στη συνέχεια, ώστε να συνεχίζονται να αναπτύσσονται πρωτοβουλίες και να μην εξαφανίζονται, να μην σταματούν. Και όπως είπε και συνάδελφος, η κυρία Τσίβλε, στη Ρήγα οι άνθρωποι που είχαν πρόσβαση στον πολιτισμό ήταν πολύ περισσότεροι μετά την πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Και αυτό ακριβώς είναι που θέλουμε να πετυχαίνουμε, να αυξήσουμε τον αριθμό των ανθρώπων που καταναλώνουν εντό εισαγωγικών πολιτισμό. Τώρα όσον αφορά την ε, ομοφοβία, ε, δεν μπορώ να δεχτώ αυτή την ιδέα ότι η βουλγαρική κοινωνία είναι έτσι. Υπάρχουν ε, οι πολιτικοί, οι οποίοι ανοιχτά το λένε ότι είναι ομοφιλόφιλοι κάποιοι τουλάχιστον. Αλλά δεν νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε τίποτα άλλο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν έχετε άλλες ερωτήσεις να κάνετε. Ε, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό τον δεύτερο γύρο ερωτήσεων που με ενέπνευσε και με συγκίνησε κιόλα. Ε, θυμάμαι πάρα πολύ καλά τις δραστηριότητες στη Ρήγα. Ε, έχω δύο ερωτήσει να υποβάλω στους ομιλητές. Επειδή ε, είσαστε όλοι εμπειρογνώμονες για την ε, οργάνωση πολιτιστικής πρωτεύουσας, ε, Πώς πιστεύετε ότι μια πρωτεύουσα μπορεί να προετοιμαστεί καλύτερα για να γίνει καλός υποψήφιος και να επιλεγεί. Και μια δεύτερη ερώτηση. Όταν επιλεγεί μια πόλη, τι θα πρέπει να κάνει έτσι ώστε να έχει αποτελεσματικό management. Πώς μπορεί να ε, συμπεριληφθεί περισσότερο η τοπική κοινωνία να συμμετέχει και αυτή πιο ενεργά στο πρόγραμμα. Πολύ ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Αν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, θα ήθελα εγώ να κάνω μία ερώτηση. Ε, τώρα πάρα πολλοί είπαν ότι σε τελική ανάλυση ε, λείπει ένα καλά οργανωμένο δίκτυο, ότι υπάρχουν άτυπες ε, συνεργασίες, ε, υπάρχουν βέβαια και επαφές ανάμεσα στις πόλεις, αλλά κατ' ουσίαν δεν υπάρχει ένα δίκτυο που να το στηρίζουν όλοι. Και νομίζω ότι αυτό κατέστη απόλυτα σαφές και κατά την τελευταία θητεία το συζητήσαμε. τι ακριβώς λοιπόν χρειάζεται αυτό το δίκτυο τι ακριβώς μπορούμε να κάνουμε κατά την άποψή σας, τι είναι απαραίτητο, πού ακριβώς ε, χρειαζόμαστε υποστήριξη και ποια είναι τα θέματα εκείνα τα οποία ε, θεωρείτε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικά αν επιθυμεί κανείς ε, να φτιάξει ένα τέτοιο δίκτυο. Έχετε συγκεκριμένες προτάσεις. Ε, θα ήθελα ε, στη συζήτηση αυτή, αν θέλετε, να συμμετέχουν όλοι ε, οι πολιτιστικές πρωτεύουσες Ρίγα και Ματέρα. Ε, για τη Ματέρα νομίζω έχουμε συζητήσει Κύριε Ταραντίνο, ε, στη Ματέρα αυτό το δίκτυο είναι κάτι το οποίο το υιοθέτησε και η ίδια η πολιτιστική πρωτεύουσα η Ματέρα. Νομίζω λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό να έρθουν κοντά όλοι οι άμεσοι ενδιαφερόμενοι ε, για να ε, είναι γνωστό το τι μπορεί να ε, φέρει ένας οργανισμός και τι μπορεί μετά να συμπληρωθεί εκ των υστέρων από μια πολιτιστική πρωτεύουσα. Αυτές είναι δύο ερωτήσεις που απευθύνονται στις δύο τελευταίες ομιλήτρες, αλλά αν θέλετε μπορείτε να απαντήσετε και άλλοι. όποιος θέλει μπορεί να παρέμβει στη συζήτηση. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να απαντήσω και στις προηγούμενες ε, ερωτήσεις. Ε, ε, θα προσπαθήσω λοιπόν να συνδυάσω όλες τις ερωτήσεις. Θα ξεκινήσω με την ιδέα του δικτύου ή κάποιας μορφής δομή που πρέπει να δημιουργηθεί. Κοιτάξτε, εγώ έχω λίγο διαφορετική άποψη. Ε, το project των πρωτευουσών ε, είναι ένα συγκεκριμένο project για μια συγκεκριμένη πόλη. Βεβαίως υπάρχουν αυτά που ονομάζουμε legacy, το κληροδότημα ή αυτά που μένουν και μετά το τέλος ε, της πολιτιστικής πρωτεύουσα, τα πράγματα που έχουμε μάθει. Ωστόσο δεν είμαι σίγουρο, σίγουρη ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί κάποια οργάνωση ή κάποια δομή ε, γιατί δεν πιστεύω ότι θα είναι ιδιαίτερος ε, εποφελές κάτι τέτοιο. Δηλαδή δεν θα προσφέρει κάτι ιδιαίτερα περισσότερο από ότι το άτυπο δίκτυο στο οποίο ε, συμμετείχαμε και ότι θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο. Στην ουσία και αυτό νομίζω ότι έχει φανεί από όλες τις παρεμβάσεις. Ε, το διαμέρισμα των εμπειριών είναι το πιο σημαντικό. Το να μοιράζεσαι εμπειρίες, να μοιράζεσαι συναισθήματα με τους άλλους. Και για να απαντήσω και στις άλλες ερωτήσεις που υποβλήθηκαν. Ναι, αναφερθήκατε ε, προηγουμένως ε, στην περίπτωση του Βλόμπερτ και ναι, το καταλαβαίνω αυτό. Η ελευθερία η ελευθερία σκέψης, η ελευθερία δημιουργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν θα πρέπει να υπάρχει κανενός είδους λογοκρισία ε, ε, να λέμε σε κάποιον αυτό δεν μπορείς να το κάνεις ή δεν μπορείς να ασκήσεις κριτική ή να είσαι επικριτικός. Ε, ακόμα και αν αυτό που κάνει είναι οδυνηρό. Ε, με τον τρόπο αυτό οθούμε και το κοινό να σκεφτεί για ορισμένα πράγματα. Σε αυτήν την περίπτωση ε, σκεφτήκαμε ε, την ελευθερία της δημιουργίας, την ελευθερία του δημιουργήν που με κανένα τρόπο δεν θα πρέπει να περιορίζεται. Όσον αφορά την ερώτηση για την πρωτοβουλία και πόσο γνωστή είναι, αν λάβω υπόψη μου την περίπτωση της ε, Ρήγας, ε, μπορώ να σας πω ότι εάν κανείς έχει περιορισμένο προϋπολογισμό, τότε θα πρέπει να σκεφτεί πολύ προσεκτικά πού θα τον δαπανίσει. Ε, και ε, στην περίπτωση της Ρήγα δεν δόθηκαν χρήματα για το μάρκετινγκ, δόθηκαν τα χρήματα για την δημιουργική διαδικασία. Και είναι αλήθεια ότι εμείς αναγκαστήκαμε να θυσιάσουμε ε, κάποια χρήματα που θεωρητικώς θα έπρεπε να δοθούν για την προώθηση και την διαφήμιση. Ε, ξέρω ότι υπάρχουν όμως άλλες ε, ε, πόλεις πολύ μεγάλες οι οποίες προβληματίζονται πολύ σχετικά με τον προϋπολογισμό που θα δώσουν και επίσης ενδεχομένως καλούνται να δημιουργήσουν οργανισμούς, φορείς για την επικοινωνία. Πάντα όμως πρέπει να γίνονται επιλογές στην ε, περίπτωση τη δική μας, εμείς επιλέξαμε την δημιουργική διαδικασία έναντι της ε, ε, πρόθεσης και της διαφήμισης. Όσον αφορά την συζήτηση για τις επενδύσεις που γίνονται στις υποδομές, υποδομές για τον πολιτισμό, υποδομές γενικά. Η, Ευρω... Ο Ευρωπαϊκός Πολι... η Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα είναι ένας συνολικό, έχει ένα συνολικό στόχο να ε, πιστούν ε, πόλεις, περιφέρειες, ακόμα και χώρες ότι θα πρέπει να δημιουργήσουν πολιτιστική υποδομή. Ωστόσο, ε, το project της πολιτιστικής πρωτεύουσας δεν είναι οικοδομικό project. Εμείς ξεκινήσαμε ε, την στιγμή της ε, κρίσης και το θέμα της υποδομής ε, δεν, ούτε καν συζητήθηκε γιατί δεν υπήρχαν κονδύλια για κάτι τέτοιο. Αλλά βλέποντας το θέμα έτσι πιο γενικά πιστεύω ότι το project των πρωτευουσών δεν θα πρέπει να βασίζεται κυρίως στην δημιουργία υποδομής. Θα πρέπει να αφορά ε, την, ε, το να πιστούν οι κεντρικές αρχές να επενδύσουν ε, στην, στον πολιτισμό και σε κάποιες υποδομές του πολιτισμού. Αυτό που θα ήθελα να πω σε άλλες ευρωπαϊκές πολιτιστικές πρωτεύουσες είναι το εξής. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι αυτό το project μπορεί να αποτελέσει ένα καλό όχημα, μια κινητήρια δύναμη για να, σε, να σου δώσει να καταλάβεις ε, τι συμβαίνει στις πόλεις ε, πολιτιστικά μιλώντας. Χρειαζόμαστε, πιστεύω εγώ, τα πέντε χρόνια αυτά για να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε, να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο δρούμε, τον τρόπο με τον οποίο ε, αντιλαμβανόμαστε τον πολιτισμό. ε, εμείς σκεφτήκαμε πάρα πολύ τι μπορούσαμε να κάνουμε σε επίπεδο πόλης, το οποίο μετά να μπορεί να μετατεθεί και σε εθνικό επίπεδο. Βεβαίως, βεβαίως ε, δημιουργήθηκαν και κάποιοι πολιτικοί συνασπισμοί και, κάποιοι, και κάποιες αντιπαλότητες και κάποιες συγκρούσεις. Ωστόσο καταφέραμε να βρούμε ε, συνενέσεις Jāsaka tā, jā, mēs visi zinām to, ka e, politiski procesa dēļ ļoti daudzās Ευρώπης κουλτούρας δάουσπιζάτας νο, νο... Νομίζω ότι αυτό πρέπει να συνέβει στις περισσότερες ε, ε, πολιτιστικές πρωτεύουσες και είναι γεγονός ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις είδαμε να αλλάζει η διοίκηση ε, στη διάρκεια της ε, διαδικασίας είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, να συζητούμε. Εμείς συζητήσαμε, καταφέραμε να πείσουμε τις αρχές για τα προγράμματα, για τα σχέδια τα οποία είχαμε. Αυτό πιστεύω ότι πρέπει να κάνουν οι πολιτιστικές πρωτεύουσες. Ευχαριστώ. Ja, vielen Dank. Ähm, okay. Πολύ ωραία. Κύριε Ταραντίνο, ευχαριστώ πολύ. Αρχίζω από την πρώτη ερώτηση. για την περίπτωση του Blogger. Και αυτή τη λογοκρισία που αναφέρθηκε. Το θετικό είναι ότι η... ο θεσμός της πολιτιστικής πρωτεύουσας ακριβώς έσπασε τις προκαταλήψεις Και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Ακούω τη φωνή μου στα ακουστικά, λέει η ομιλήτρια και δυσκολεύομαι. Λοιπόν, ε, από την άλλη μεριά, βέβαια, στα μέσα ενημέρωση με ανακοινώσει. Στηρίχθηκε το Πλόντιφ. Αλλά είναι κάτι που συζητήσαμε όταν είχαμε μια οικογενειακή συνάντηση, ας πούμε, για τα καλλιτεχνικά, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και ο Ξαβιέ το έθεσε. Το κατά πόσο δηλαδή θα πρέπει να γίνεται πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης, μια πόλη η οποία δεν σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όντως είναι ένα ζήτημα που τίθεται. Πάντως χαρικά πάρα πολύ στον πλότο πραγματικά πέρασα πάρα πολύ ωραία και ήμουν ενθουσιασμένη που μπόρεσα να συνεργαστώ με ανθρώπους που είχαν τόσο ανοιχτό πνεύμα. Η συνεργασία μας ήταν πάρα πολύ καλή και τους θαυμάζω που τολμούν για το θάρρος τους. Ακριβώς, γιατί είναι πολύ θαραλέοι και κατάφεραν να κάνουν και αυτή την έκθεση που έκαναν. Έρχομαι τώρα στο θέμα της ματέρα. Όντως, έχουμε κρατήσει μια κληρονομιά από όλη αυτή την ιστορία. Ε, θα οργανώσουμε κάτι και είσαστε όλοι προσκεκλημένοι βέβαια. Και με άλλες πολιτιστικές πρωτεύουσες θέλουν να ετοιμάσουμε κάτι και να το δώσουμε στον κύριο Σασόλη όταν έρθει στη Ματέρα στις 20 Δεκεμβρίου. Ευχαριστώ να έχουμε και εσάς. Και η πρόσβαση για μας είναι κάτι πολύ σημαντικό. Γιατί χρησιμοποιούμε ένα πάσο, μια κάρτα, η οποία δίνει πρόσβαση στα πάντα, σε όλες τις εκδηλώσεις, μικρές, μεγάλες, εργαστήρια. και οποιασδήποτε ηλικία άνθρωποι, όλοι μπορούν να συμμετέχουν ε, σε αυτές τις διαδρομές. Τώρα για την Ευρωπαϊκή πολιτιστική πρωτεύουσα για το θεσμό. Αυτό που πιστεύω ότι είναι επίσης πολύ σημαντικό είναι το εξή. Πρέπει κανείς να ξανασκέφτεται την πόλη, να την ξαναγεννάει. Αν έχετε να δουλέψετε πάνω σε αυτό το θεσμό, να ξέρετε ότι είναι μια τεράστια ευκαιρία και ότι δεν δουλεύετε μόνο με τους τοπικούς παράγοντες και τον κόσμο επιτόπου, αλλά και με εξωτερικούς παράγοντες γιατί μπορεί αυτοί να δούνε κάτι που εσείς δεν βλέπετε που σας τα πω μέσα. Οπότε δεν είναι ένα τοπικό εγχείρημα θα έλεγα εγώ. Δεν θα έπρεπε. Και χρειάζεται και στενή συνεργασία με τους πολίτες, με τους θεσμούς, γιατί οι θεσμοί θα σας δώσουν τη στήριξη για να κάνετε πράγματα. Οπότε πρέπει να έχετε αυτή τη στήριξη και από την άλλη μεριά με τον κόσμο, γιατί ο κόσμος σας δίνει τη μεγάλη ευκαιρία να φτάσετε σε αυτόν. Για το θέμα της δικτύωσης. Πιστεύω, και εδώ θέλω να επανέλθω στο θέμα της επικοινωνίας, το δίκτυο έχει, δίνει πολλές δυνατότητες. Ενισχύει την επικοινωνία μαθαίνονται πολύ περισσότερα πράγματα μέσω ενό δικτύου για την πολιτιστική πρωτεύουσα, γιατί μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους πόρους μας, μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερο αντίκτυπο στην ε, επικοινωνία. Αυτό δηλαδή δεν είναι θέμα της ματέρα μόνο, είναι ευρωπαϊκή υπόθεση, είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα και έτσι πρέπει να προβάλλεται. Πρέπει να έχει λοιπόν αντίκτυπο ευρωπαϊκό οτιδήποτε γίνεται. Και ένα παράδειγμα μπορεί να μην είναι πολύ σημαντικό, αλλά εμείς έχουμε web team, δηλαδή ομάδες που είναι εθελοντές και βοηθούν ε, να περνάμε στο διαδίκτυο πράγματα για την πολιτιστική μας πρωτεύουσα. Αυτούς θα μπορούσαμε να τους ανταλλάξουμε, για παράδειγμα, μεταξύ μας. Θέλω να πω ότι υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να κάνουμε μαζί και μία στο σελίδα μπορεί να μιλάει και για άλλα πράγματα, όχι μόνο για την τρέχουσα πολιτιστική πρωτεύουσα, αλλά και για τις προηγούμενες και για τις επόμενες και να εξηγεί τι γίνεται όχι μόνο στις μεγάλες πόλεις, αλλά και στις μικρές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδοτεί τώρα μία πρωτοβουλία για να βοηθήσει τις επόμενες πολιτιστικές πρωτεύουσες για να υπάρξουν και δραστηριότητες δικτύωσης. Πάντως, αυτά τα δίκτυα θα έπρεπε να ενισχυθούν, να προωθηθούν, κατά τη γνώμη μου. Και υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε μαζί, είτε υπέρ του τουρισμού, μείωση της γραφειοκρατίας, οικοδόμηση ικανοτήτων κλπ. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ. Μία απάντηση από εδώ. Ναι, παρακαλώ. Θέλω να αντιδράσω σε δύο πράγματα. Πρώτον, ε, σε σχέση με το δίκτυο, είχα την εντύπωση ότι θα είμαι στη μειονότητα, αλλά πρέπει να σας πω ότι υποστηρίζω πλήρως ε, ε, το ότι θα πρέπει να διατηρηθεί αυτό το δίκτυο εφόσον υπάρχει. Το μέλλον ε, δείχνει ότι θα πρέπει να φιλοξενήσουμε και άλλες πολιτιστικές πρωτεύουσε. Ε, δεν υπάρχει καμία γραφειοκρατία, δεν υπάρχει τίποτα, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο για να μπορεί κανείς να αποφεληθεί από αυτό το άτυπο δίκτυο. Ε, εγώ ήμουνα κατά του να είναι μια επίσημη πλατφόρμα κάτω από το Creative Europe, αλλά ο Σιλβάν Πασκουάρ που είναι αρμόδιος για την επιλογή. Εκείνος βέβαια μπορεί να σας ενημερώσει πολύ καλύτερα για το επίσημο δίκτυο που είναι ένα δίκτυο ε, δημιουργίας ικανοτήτων για τις ε, μελλοντικέ ε, πολιτιστικές πρωτεύουσες. Αυτό φτάνει για μένα, είναι πολύ καλά οργανωμένο. Και τώρα μία πολύ σύντομη αντίδραση στο θέμα του Plovdiv και της Βαλέτα. Πριν από λίγο αναφέρατε ότι με κάθε σεβασμό για αυτά που συνέβησαν στο Plovdiv Τελικά όμως ε, το όλο θέμα στέφτηκε από επιτυχία. Ήταν μια μεγάλη δυσκολία για την ομάδα, τα κατάφεραν, επιβίωσαν, ε, διαφύλαξαν το κύρος τους, ε, οργανώθηκε και η εκδήλωση στην εποχή του λαϊκισμού και της δύναμης της ισχύω των μέσων ενημέρωσης. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να συμβεί παντού. Ένας λαϊκιστής πολιτικός να θέσει ένα θέμα και στο Πλόβδιβ ε, τελικά ε, κατόρθωσαν να το ξεπεράσουν. Ε, τώρα, αυτά που συνέβησαν στη Βαλέτα για μένα είναι τελείως διαφορετικά, παντελώς απαράδεκτα και εγώ δεν βλέπω καμία επιτυχία σε αυτή την ιστορία της λογοκρισίας, του να κρύβει κανείς γεγονότα, εγκλήματα και όλα τα σχετικά και δυστυχώς ε, δεν υπάρχουν εργαλεία για να γίνουν βήματα κατά τέτοιων περιπτώσεων πολιτιστικών ε, πρωτευουσών. Ε, νομίζω ότι η Επιτροπή δεν μπορεί να κάνει τίποτα δεν μπορεί να κάνει τίποτα σε διοικητικό επίπεδο. Βεβαίως μπορούν να γίνουν κάποια βήματα από τους πολιτικούς. Ξέρω ότι πάρα πολλοί αρνήθηκαν να πάνε στην τελετή έναρξης αυτό ως διαμαρτυρία. Ε, κατά των πολιτικών, υψηλόβαθμων πολιτικών. Τώρα δεν θυμάμαι πόσο στεναρή ήταν η αντίδραση των πολιτικών, πάντως εγώ θα την ήθελα ακόμα πιο στεναρή. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, είναι δύσκολο να μιλήσει κανείς μετά τον προλαλήσαντα, γιατί με κάλυψε. Είπε αυτά που θέλω να πω. Και εγώ θέλω να πω ότι το δίκτυο θα ήθελα να παραμείνει ως έχει. Είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό και αν ήταν επίσημο θα ήταν δύσκολο να μπορεί κανείς ε, να ε, ορίζεται το ποιος θα είναι μέλος και ποιος όχι. Ε, ποιος θα είναι μέλος, θα είναι οι πόλεις, θα είναι οι άμεσα εμπλεκόμενοι και ενδιαφερόμενοι. Έτσι λοιπόν, κάτω από αυτή τη διάσταση του θέματος, το δίκτυο θα μπορούσε να μετατραπεί σε ένα ε, επίσημο δίκτυο όπου θα συμμετέχει ο Δήμαρχος και διάφοροι άλλοι, αλλά τότε πια δεν θα είναι ε, λειτουργικό, ε, θα γίνει ένα βαρετό δίκτυο σαν αυτά που ξέρουμε να υπάρχουν πολλά στην Ευρώπη, παντελώς βεριτά, βαρετά. Και αυτό θα ήταν μεγάλη απώλεια. Κατά τα άλλα υπάρχουν βέβαια καθήκοντα και πράγματα τα οποία συζητάμε συνεχώς. Ίσως τώρα να μην είναι ιδιαίτερα επίκαιρα, αλλά παρήματο χάρη το θέμα ενός αρχείου. Δηλαδή ε, όλη αυτή τη γνώση και την εμπειρία, πώς μπορεί κανείς να τη μεταφέρει πιο κάτω. Ε, κατά την άποψή μου, με την ψηφιοποίηση μπορεί κανείς να πετύχει πάρα πολλά, όχι τα πάντα, αλλά πολλά. Και γι' αυτό αυτός ο χαρακτήρας ε, του δικτύου που μοιάζει με διάλογο είναι πολύ χρήσιμος. Μπορούμε να ε, μεταδώσουμε αυτά που δεν αναφέρονται και δεν περιλαμβάνονται στο διαδίκτυο. Είπα ότι μερικές φορές ε, αναζητάμε περαιτέρω δυνατότητες για το δίκτυο. Στη Μάλτα, παραδείγματο χάρη, θα θυμάστε ίσως, είχαμε μία περίπτωση όπου από την πολιτιστική πρωτεύουσα υπήρξαν κάποιες δηλώσεις για την δολοφονωμένη δημοσιογράφο, για την οικογένειά της, που ήταν παντελώς απαράδεκτες. Εμείς λοιπόν συντάξαμε μια επιστολή και τη στείλαμε. Περισσότερα δεν μπορούμε να κάνουμε αλλά τέτοιου είδου συμβολικέ χειρονομίε νομίζω ότι είναι σημαντικέ. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει τίποτα παραπάνω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριο Ρουΐσε. και μετά πρέπει να αλλάξουμε το πάνελ γιατί έχουμε άλλους τρεις ομιλητές και δεν ε, έχουμε εδώ χώρο για να τους φιλοξενήσουμε όλους. Ευχαριστώ. Ποιος ε, κοιτάει τις 60 σελίδες στην ιστοσελίδα αν υπήρχε ένα δίκτυο, τότε θα υπήρχαν σε αυτό το δίκτυο αυτές οι σελίδες των πολιτιστικών πρωτεύουσών. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να ανοίξει η συζήτηση, δηλαδή πώς να είναι αυτό το δίκτυο. Δεν ξέρω αν καλύτερα με αυτόν ή τον άλλο τρόπο. Πάντως, στην Επιτροπή Πολιτισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα μπορούσε κάλλιστα πάλι καλά εδώ, αλλά θα μπορούσε και σε άλλο επίπεδο. Υπάρχουν πράγματα πάντως γραπτά, τα οποία θα μπορούσαν να μελετηθούν. Δεύτερον, για τα πέντε χρόνια, αν κάποιος μπορεί να μου πει εδώ πού πρέπει να βρίσκεται ο ευρωπαϊκός πολιτισμός σε πέντε χρόνια και το πετύχει, ε, τότε σημαίνει ότι δεν έχουμε προχωρήσει αρκετά. Θα μπορούσαμε να είχαμε προχωρήσει περισσότερο. Πέντε χρόνια είναι πολλά αλλά και λίγα. Το περιθώριο σφάλματος πάντως και οι προοπτικές για τις πόλεις που είναι υποψήφιες καλύτερα ταιριάζουν τα τρία χρόνια. Και τέλος συμφωνώ με ότι είπαν οι συνάδελφοι από τις πολιτιστικές πρωτεύουσε για το ανθρώπινο δυναμικό. Τα ανθρώπινα δικαιώματα πράγματι είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθούμε μαζί, αλλιώς δεν θα πάμε πουθενά. Πολλά χρόνια πολύ πολύ ύπνο έχω χάσει, αλλά να ξέρετε ότι είμαι πολύ ευτυχισμένος που ασχολήθηκα με τις πολιτιστικές πρωτεύουσες Ευρώπης. Θα ήθελα τώρα να παρακαλέσω να γίνει γρήγορα η αλλαγή ε, στο πάνελ για να συνεχίσουμε με το δεύτερο γύρο. Και ευχαριστώ όλους εκείνους που ήρθαν σήμερα και που μας παρουσίασαν μια πολύ ενδιαφέρουσα άποψη για το θέμα των πολιτιστικών πρωτευουσών. Για μας έχει πολύ ενδιαφέρον να ακούμε ε, από την πρακτική εφαρμογή ανθρώπους που τα έζησαν όλα αυτά και νομίζω ότι ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα ακρόαση για όλους μας ε, και έχουμε τώρα τους εμπειρογνώμονες. Ε, θα ακούσουμε τώρα τη δική τους άποψη. und ich darf äh, Frau Ammann, äh, Frau Blase und äh, Frau Ammann, Blase και Garcia ε, θα ήθελα να καλέσω παρακαλώ να έρθετε εδώ να καθίσετε στο βήμα. Ja, ich glaube, hier oben hat jetzt jeder soweit Platz genommen. Παρακαλώ να καθίσετε. Moment, hier fehlt der, der, der. Maybe at the very end. At the very end, yeah. yeah. und ich darf... Και όπως σας είπα, θα ήθελα να καλωσορίσω εδώ στο βήμα την κυρία Αμάν και η κυρία Μπλάζερ που έχουν από κοινού 5 λεπτά και μετά η κυρία Γκαρσία έχει άλλα 5 λεπτά. Και θα ήθελα να παρακαλέσω τώρα να τηρήσουμε λιγάκι το χρόνο. Ξέρω ότι ε, έχουμε καθυστερήσει λιγάκι, αλλά θέλουμε μετά να ακολουθήσει και διάλογος. Αυτά τα οποία δεν ελέγχθησαν ή δεν θα υποθούν στην αρχή, ε, μπορούν να υποθούν μετά στις ε, ερωταπαντήσεις. Παρακαλώ, κυρία μας. Yes, thank you very much for inviting us. Um, so we will do our presentation. Ευχαριστώ πολύ. Θα κάνουμε μαζί ε, την παρουσίασή μας ε, με την Αγνιέσκα. Πριν από πέντε χρόνια εμείς είμαστε στο κοινοβούλιο εδώ στο πάνελ ε, και ξεκινήσαμε πολύ κοινή δουλειά, συνεργατική και ε, γι' αυτό θεωρήσαμε ότι θα έπρεπε και οι δύο να κάνουμε την παρουσίαση. Θα μιλήσουμε λοιπόν για τον τρόπο με τον οποίο καλύτερα μπορούμε, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ε, το πλήρες δυναμικό των ευρωπαϊκών πολιτιστικών ε, πρωτευουσών. Θα δώσουμε και κάποιες σκέψεις για μελλοντικές βελτιώσεις ε, είναι γεγονός ότι είναι επιτυχημένη πρωτοβουλία αυτή των ε, πολιτιστικών ε, πρωτεύουσών από πολλές πλευρές και προοπτικές. Ο ρόλος μας εδώ στο πάνελ ίσως είναι, στο πάνελ εδώ είναι ίσως να σας δείξουμε και τι συμβαίνει αλλά και τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον. Ξέρουμε και βλέπουμε ότι υπάρχει ε, μεγάλο ενδιαφέρον εντός και εκτός ακόμα της Ευρώπης. Αποτελεί πηγή έμπνευσης αυτή η ιδέα ε, και ο θεσμός των πρωτευουσών. Ε, υπάρχει πολύ δυναμικό, πολλές νέες ευκαιρίες και νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε από αυτήν την ιδέα έτσι ώστε να προχωρήσουμε παραπέρα. Πολλά μπορούν, έχουμε να πούμε θα προσπαθήσουμε να σκιαγραφίσουμε τα κεντρικά στοιχεία. Θα ήθελα βέβαια να πω ότι και οι δύο οριστήκαμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά υπάρχει και η Χριστίνα Φερένια, η συνάδελφός μας. Είμαστε τρεις γυναίκες λοιπόν που ε, εσείς επιλέξατε. Και αυτό έφερε και την ε, διαφοροποίηση του φύλου. Θέλαμε να το υπογραμμίσουμε και αυτό ως στοιχείο. Πιστεύω ότι ε, μπορούμε να πούμε ότι δουλέψαμε ε, με δύο, βασιζόμενοι σε δύο αρχές. Πρώτα, προσπαθήσαμε να βρούμε τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα ε, στις χώρες και ε, ε, βεβαίως εμείς έχουμε και την υποχρέωση του, της επιτήρησης, παρακολούθησης, του monitoring. Αυτή τη στιγμή έχουμε 10 διεθνείς ε, ε, εμπειρογνώμονες με δυνατότητα να προσθεθούν και δύο εθνικοί εμπειρογνώμονες άρα υπάρχει πολυμορφία όσον αφορά την ε, πραγματογνωμοσύνη ακολουθούμε πέρα από την ε, ισορροπία των φύλων ακολουθούμε και ένα δημοκρατικό ε, πλαίσιο ε, εργασίας. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε αυτό το brand των ευρωπαϊκών πρωτευουσών με ταυτόχρονη διατήρηση της ποιότητας των προγραμμάτων. Επίσης πιστεύω ότι αυτό που είναι σημαντικό να πούμε εδώ είναι ότι έχουμε πολλά παραδείγματα πάρει από προηγούμενες πολιτιστικές πρωτεύουσες, αλλά τώρα βρισκόμαστε σε ένα σημείο καμπής, ε, γιατί από του χρόνου οι νέοι κανόνες ε, θα αρχίσουν να εφαρμόζονται. Ε, γι' αυτό εδώ έχουμε βάλει το νέο χρονοδιάγραμμα των πολιτιστικών πρωτεύουσών, ε, φτάνουμε μέχρι την ε, Γερμανία και τη Σλοβενία που, είναι, που συμμετέχουν ε, στο, στο, διαγωνισμό ως υποψήφιες είναι ανάγκη να καταλάβετε εκ των προτείνων ότι αλλάζουν οι προϋποθέσεις σε σχέση με αυτό και το πλαίσιο σε σχέση με αυτό που είχαμε μέχρι τώρα. Εδώ βλέπετε έξι κριτήρια τα οποία εμείς έχουμε επιλέξει για τις νέες ε, ε, πρωτεύουσες από το 20 μέχρι το 33. Ε, και θα θέλαμε να αναφερθούμε σε ορισμένα από αυτά. Ας πούμε, ε, μακροχρόνια στρατηγική ε, και legacy. Στο προηγούμενο πλαίσιο υπήρχαν μονάχα δύο κριτήρια και αυτά όχι σαφώς καταγεγραμμένα. Εδώ υπάρχουν έξι πλέον κριτήρια με διάφορες κατηγορίες υποκριτηρίων σε ένα πολύ διαρθρωμένο δομημένο πλαίσιο όσον αφορά τις βελτιώσεις, τι θα μπορούσε δηλαδή να γίνει με καλύτερο τρόπο. Εδώ αναφέρονται πολλά στοιχεία, εγώ θα αναφερθώ μονάχα σε δύο. Πιστεύω ότι όλο και περισσότερο γίνεται κατανοητό ότι η πόλη δεν είναι κάτι εξωεδαφικό. Ε, είναι ένα ε, ε, έδαφος το οποίο περιβάλλεται από την περιφέρεια. Ε, και επομένως πιστεύουμε ότι θα πρέπει να ε, διαγωνίζονται οι πόλεις μαζί με την περιφέρεια έτσι ώστε να υπάρχει συνεκτική προσέγγιση ισχυρή μάλιστα συνεκτική προσέγγιση. Επίσης αυτό που αναφέρθηκε ήδη και προηγουμένως ε, και είναι πολύ σημαντικό είναι η δημοσιονομική σταθερότητα, η σταθερότητα όσον αφορά τον προϋπολογισμό γιατί ακόμα ο ίδιος ο τίτλος της ε, πολιτιστικής πρωτεύουσας, ε, ακόμα και για μικρές πόλεις, μπορεί να δημιουργήσει ε, ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα μόχλευσης και ε, επομένως ε, μπορεί να υπάρξουν και συνδιαχειρήσεις ή ε, πολυεπίπεδη διαχείριση κτλ. Από την άλλη πλευρά βέβαια αυτό είναι πιο δύσκολο γιατί αναφέρθηκε κιόλας και το είδαμε ότι μερικές φορές οι προσδοκίες ή μάλλον οι δεσμεύσει δεν ολοκληρώθηκαν και επομένως αυτό μπορεί να βαραίνει πάρα πολύ στην προετοιμασία του έτος γιατί εάν δεν υπάρχει το απαραίτητο χρηματικό χρηματοδοτικό πλαίσιο έτσι όπως το είχες αρχικά ε, καθορίσει, προφανώς ε, δεν μπορεί να συνεχίσει να προωθηθεί καλά η δουλειά. Ε, και επίσης πρέπει να υπάρχει δυνατότητα για επιπλέον προσωπικό, για δραστηριότητες προσέγγισης, μεγαλύτερης προσέγγισης, outreach activities. Επίσης, σε γενικές γραμμές, κατά τη δική μας άποψη, ε, όλη η χώρα ε, μπορεί να επωφεληθεί από την ε, ε, πολιτιστική πρωτεύουσα. Άρα θα πρέπει να συμμετέχει με κάποιο τρόπο. Οι νέοι κανόνες ε, μάλιστα αναφέρονται ε, συγκεκριμένα και σε πολιτιστική βελτίωση, πολιτιστικά πλεονεκτήματα και επομένως θα πρέπει έτσι να το δουν και οι χώρες και όχι μονάχα σε έναν διαγωνισμό εξειδικευμένο για την πόλη. Επομένως, η πολιτιστική πρωτεύουσα δεν αφορά μονάχα την ίδια την πρωτεύουσα, αλλά ε, την ε, και την συνεργασία και την ανάπτυξη και την διαφοροποιημένη συνεργασία με διάφορους ε, παίκτε. επίσης, αφορά την επένδυση στην capacity building, οικοδόμηση ικανοτήτων, όχι μονάχα όμως στον πολιτισμό, αλλά γενικά. Αφορά επίσης την συμμετοχή των πολιτών, όχι μονάχα σε τοπικό επίπεδο αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ένα από τα θετικά στοιχεία για το θεσμό των πολιτιστικών πρωτευουσών είναι ο αντίκτυπος που μπορεί να έχουν στις πόλεις που τώρα είναι πλέον μεγαλύτερος. Ε, η κοινωνική συνοχή είναι ένα από τα ζητήματα τα οποία ιδιαίτερως υπογραμμίζουμε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μας. Και τώρα φτάνουμε ε, στο κεντρικότερο στοιχείο. Ακούσαμε πολλά για την πολιτιστική ανάπτυξη των πόλεων, αλλά η πραγματική ε, διαφοροποίηση από τοπικό, περιφερειακό, εθνικό επίπεδο ε, πολιτισμού είναι ότι στην ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, πολιτιστική πρωτεύουσα, έχουμε ακριβώς την ευρωπαϊκή διάσταση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε και το στοιχείο αυτό και ε, οι πολιτιστικές πρωτεύουσες είναι μία, αν όχι η κεντρικότερη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι γνωστή, που γίνεται γνωστή σε όλο τον κόσμο, που είναι ορατή από όλους σε ε, παγκόσμιο επίπεδο ε, και επομένως εξαρτάται, ε, εδώ παίζεται μάλλον, διακυβεύεται και ο τρόπος με τον οποίο θέλει η Ευρώπη να ε, γίνεται αντιληπτή από το εξωτερικό. Επίσης, η ε, προσέγγιση ε, μέσω της επικοινωνίας είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, αναφέρθηκε και προηγουμένως. Οι επιλεγμένες ε, πόλεις ε, επιλέγουν κάποια στρατηγική, υπεύθυνου στρατηγικής. Βεβαίως αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο για τις μικρές πόλεις και πρέπει όμως να γίνεται. Υπάρχει τεράστιο δυναμικό το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνέργεια και με τα ευρωπαϊκού επίπεδου εργαλεία επικοινωνίας, έτσι ώστε οι πολιτιστικές πρωτεύουσε να γίνονται πιο ορατές. Το άλλο θέμα είναι το περιεχόμενο. Αυτό το αυτή η κατανόηση της βιωσιμότητας ε, που νομίζω ότι ε, πλέον είναι μια αντίληψη που όλοι την ε, έχουμε. Ε, και αναφερόμαστε σε μια συνολική ε, αντίληψη της, ε, βιο, της βιωσιμότητας που είναι και οικονομική και πολιτιστική και, και περιβαλλοντική. Έχουμε επίσης εδώ το θέμα του τουρισμού και του υπερτουρισμού γιατί έχουμε τουρίστες που έρχονται από όλα τα μέρη του κόσμου. Το πάνελ θεωρεί ότι οι πολιτιστικές πρωτεύουσες ε, πρέπει να είναι ένα κοινό project και δεν ελέγχουμε, ε, ε, κάνουμε coaching, υποστηρίζουμε, βοηθάμε, έχουμε αυτόν τον υποβοηθητικό ρόλο και πραγματικά μέσα από αυτόν τον θεσμό μπορείτε να ενισχύσετε τον ίδιο το θεσμό και το θεσμό ανάμεσα στο τοπικό και το ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστούμε πολύ. Μακάρι να είχαμε περισσότερο χρόνο. Να τηρείτε το χρόνο σας. Πέντε λεπτά γιατί εσείς πήρατε το διπλό. Παρακαλώ, κύριε Γκαρσία. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Πολύ χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ μαζί σας σήμερα το απόγευμα. Καλησπέρα σε όλους. Θα μιλήσω ισπανικά λίγο, αλλά μετά στα αγγλικά. Πέντε λεπτά μου είπαν ότι έχω στη διάθεσή μου. Οπότε, τι θα κάνω. Θα σας πω ότι υπάρχουν πολλά στοιχεία και μεγάλη τεκμηρίωση. Εγώ είμαι διευθύντρια του παρατηρητηρίου για τις πόλεις του πολιτισμού, ερευνήτρια. Και συγκεντρώνω πληροφορίες για τις πόλεις όπου υπήρξε κάποια πολιτιστική παρέμβαση. Γιατί υπάρχουν πολιτιστικέ πρωτεύουσε τη Ευρώπη, αλλά ξέρετε ότι υπάρχουν και άλλε δραστηριότητε που εμπνεύστηκαν από το θεσμό αυτό. Οπότε εγώ έχω συγκεντρώσει πολλά στοιχεία από διάφορες πολιτιστικέ εκδηλώσεις αλλά και από άλλες όπως είναι Ολυμπιακοί αγώνε που έχουν άλλο βέβαια στόχο και πλαίσιο αλλά που αλληλεπιδρούν για κάποια πράγματα με τις πολιτιστικές πρωτεύουσε. Και είμαι επίσης μέλος της Επιτροπής που επιλέγει τις πολιτιστικές πρωτεύουσε. Το 2012 ορίστηκα με διαγωνισμό από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να εκπονήσω αυτή τη μελέτη. Είναι μια μελέτη που καλύπτει τα πρώτα 30 χρόνια του προγράμματος. Από το 1985 λοιπόν μέχρι το 2019 συγκέντρωσα στοιχεία. Ότι δηλαδή υπήρχε διαθέσιμο, ότι είχε δημοσιευθεί, ότι είχε κυκλοφορήσει για τις 60 περίπου πόλεις ε, στις οποίες ε, αναφερθήκαμε. Υπάρχουν λοιπόν βουνά τεκμηρίωσης και πληροφοριών. Το θέμα είναι πώς να βγάλουμε κάποιο νόημα από όλη αυτή την τεκμηρίωση. Εξού και εκπώνησε αυτή την μελέτη. Υπάρχουν κάποια αντίτυπα εδώ που κυκλοφορούν. Οπότε φτιάξαμε, χαρτογραφήσαμε κατά κάποιο τρόπο την κατάσταση και προσπαθούσαμε να δούμε τι είναι συγκρίσιμο και τι δεν είναι. Και αυτό που είναι πολύ χρήσιμο είναι να θυμόμαστε την ποικιλομορφία των πόλεων και των τοποθεσιών που ορίστηκαν σαν πολιτιστικές πρωτεύουσες. Γιατί αυτό το οποίο με κάνει να βλέπω τη διαφορά είναι ότι σε αντίθεση με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, εδώ εμείς την πολιτιστική πρωτεύουσα έχουμε τόσο διαφορετικές πόλεις σε μέγεθος, σε γεωγραφική θέση, στην θέση τους εθνικά αλλά και πανευρωπαϊκά. Επίσης εδώ βλέπετε πόσο διαφορετικό περιβάλλον είναι αυτό μέσα στο οποίο λειτουργήσαν οι πολιτιστικές πρωτεύουσες. Έχετε εδώ διάφορα παραδείγματα, όλα αυτά υπάρχουν γραπτά και μπορείτε να τα δείτε λεπτομερώς αργότερα. Πάντως, λίγα πράγματα που πιστεύω ότι είναι πολύ χρήσιμα. Πριν περάσουμε στα επόμενα βήματα που μοιράστηκαν μαζί μας ε, η Ανιέσκα και η Σίλβια. Εδώ. Τι πετύχαμε τα πρώτα 30 χρόνια. Με την ομάδα μου προσπαθούμε να δούμε αν υπήρξε κάποια κίνηση προς τα μπρος. Αν δηλαδή ξεκίνησε μια διαδικασία εκμάθησης, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε ένα όραμα για την πόλη που να το κάνουμε στρατηγική. Πώς συνδέεται δηλαδή για να καταλήξει σε ένα πρόγραμμα εργασίας στη συνέχεια που θα έχει κάποιον αντίκτυπο. Αυτά λοιπόν τα δοκιμάσαμε στις 60 πόλεις και εντοπίσαμε αυτές ε, τις ε, σχέσεις που βλέπετε εδώ. Θα μπορούσε κανείς βέβαια να πει περισσότερο για το τι δεν έχουμε στη διάθεσή μας και τι άλλες ερωτήσεις θα έπρεπε να κάνουμε για να έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Πάντως φάνηκε ότι να έχει κανείς ένα όραμα ε, για να αλλάξει την πόλη είναι κάτι που χρησιμοποιήθηκε πάρα πολύ στα πρώτα στάδια του προγράμματος που υπήρχε κενό. Τώρα υπάρξει τεράστια πρόοδος και βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές εξελίξεις. Ένα άλλο βασικό στοιχείο που αναπτύχθηκε και είναι ένα επίτευγμα είναι η τυποποίηση της ιδέας ότι ο πολιτισμός τοποθετείται εγκάρσια. Ότι έχει να κάνει με την ε, εκπαίδευση με την πολιτιστική κληρονομιά, αλλά ακόμη και με τις μεταφορές και τα εξηγούμε αυτά στην έκθεση. Έπειτα η λειτουργία αναθέματα ήταν κάτι πολύ σημαντικό, όπως επίσης άλλο επίτευγμα είναι ο συνδυασμός της εικόνας με τα υπόλοιπα με την δουλειά που κάνουμε συνήθως στα πολιτιστικά. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες για τα αποτελέσματα της έρευνάς μου. Πάντως, τα έγγραφα που δημοσιεύτηκαν τόσο στην έκθεση όσο και σε άλλες περιπτώσεις, όπως το Liverpool που εγώ δραστηριοποιούμε και όπου εδώ και 15 χρόνια κάνουμε την έρευνά μας, βλέπουμε πώς αυτές οι πρωτοβουλίες μπορούν να τροποποιήσουν την πολιτιστική μορφή μιας πόλης. Τα πάνε και οι συνάδελφοι αλλά και εγώ έχω συγκεντρώσει στοιχεία που δείχνουν πώς όλα αυτά γίνονται πραγματικότητα, πώς άλλαξαν οι πόλεις, από πού ξεκίνησαν, πού έφτασαν, εξαρτάται βέβαια πάντα από το σημείο κίνησης, πώς λειτουργήσαν τα δίκτυα, αν υπήρξε δυνατότητα να ξεκινήσει και να συνεχιστεί η δουλειά που ξεκίνησε με τις πολιτιστικές πρωτεύουσε. Πάντως έχουν συγκεντρωθεί στοιχεία που δείχνουν ότι είναι δυνατή μια τεράστια αλλαγή, όπως στη Λασκόβη, για παράδειγμα και στη Ματέρα. Είδαμε ότι ο θεσμός αυτός μπορεί να αλλάξει πάρα πολύ μια πόλη, η οποία μερικές φορές ξεκινάει να έχει ακόμα και κακή φήμη και μετά αποκτάει άλλο πρόσωπο. Υπάρχουν βέβαια και πολλές προκλήσεις. Στατιστικά δεδομένα υπάρχουν που δείχνουν οι τοπικές κοινότητες μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο ε, αντιμετωπίζουν οι πολίτες της πόλης τους. Εδώ βλέπουμε ότι 50-50% του τοπικού πληθυσμού νιώθει ότι έγινε καλύτερη πόλη τους. Είναι σημαντικό βέβαια να λάβουμε υπόψη μας ότι αλλάζει και το κοινό που παρακολουθεί τα πολιτιστικά δρόμενα. Μια άλλη σύγκριση που είναι ενδιαφέρουσα είναι αυτή. Δεν πρέπει βέβαια να συγκρίνουμε μήλα με αχλάδια. Οι, οι πόλεις είναι διαφορετικές μεταξύ τους και πρέπει να το έχουμε υπόψη μας αυτό. Αλλού έχουμε 30.000 επισκέπτες, ε, για κάποιες πόλεις είναι τεράστιο επίτευγμα, ε, για άλλες το 1 εκατομμύριο μπορεί να είναι ένα μέτριο αποτέλεσμα και έπειτα και οικονομικά, όπως υπόθηκε και πριν, υπήρξε μεγάλη πίεση για τα οικονομικά αποτελέσματα. Νομίζω ότι είναι σημαντικά βέβαια, αλλά δεν είναι ε, το μόνο κριτήριο που πρέπει να μας οδηγεί στο συμπέρασμα το αν κάτι πήγε καλά ή όχι. Έχουμε, όπως σας είπα λοιπόν, πάρα πολλά στοιχεία, αλλά όλα αυτά τα στοιχεία της καλλιώς πρέπει κανείς να τα βάζει στο σωστό πλαίσιο. Από πλευράς τουρισμού πάντως πρέπει να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουν οι πόλεις το ρυθμό του τουρισμού και να καταλάβουν επίσης ότι όταν έχουν πάρα πολύ τουρισμό κάποια στιγμή, ε, κάποια άλλη στιγμή έχουν και πολύ χαμηλά επίπεδα τουρισμού, κάτι το οποίο με το χρόνο μπορεί να είναι μια δυσκολία. Όλα αυτά τα αφήνω σαν τροφή για σκέψη. Υπάρχει το υλικό και online να ξέρετε και τα γραφήματα, αλλά υπάρχουν και παραρτήματα με λεπτομέρειες, με πληροφορίες που σίγουρα θα μπορούσαν να βοηθήσουν πολύ, ενημερωτικά δηλαδή για τις διάφορες πόλεις, πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης. Αυτά είχα να σας πω σήμερα και ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, κάτι να ρωτήσω αυτή η μελέτη είναι του 2013. Υπάρχουν ε, προσθήκες ε, σε αυτή τη μελέτη που να ε, περιλαμβάνουν πιο επίκαιρα στοιχεία, γιατί έχουν περάσει έξι χρόνια και ίσως να έχει αλλάξει το μεταξύ και ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζονται οι πολιτιστικές πρωτεύουσε. Μικρόφωνο παρακαλούμε. πάρα πολύ σημαντική αυτή η ερώτηση. Ως ακαδημαϊκός και κάποιος ε, που αξιολογεί το θέμα του χρόνου, είναι σημαντικό πώς προκύπτουν οι εξελίξεις. Η αξία αυτής της ε, μελέτης είναι ότι εξετάζει τα δεδομένα σε ένα χρονικό διάστημα 30-33 ετών. Ε, η δουλειά που κάνουμε συνεχίζεται και αυτό που βασικά είναι η δουλειά μας είναι να εντάσσουμε στο σύστημα τα στοιχεία, δηλαδή συμπληρώνουμε με πληροφορίες. Και ε, το θέμα είναι πώς τα επικοινωνούμε όλα αυτά. Ε, έρχονται οι πληροφορίες, έχουμε τις ε, μεθόδους ε, και τις τεχνικές. Βεβαίως είναι πολύ ενδιαφέρον το τι θα γίνει με την οικοδόμηση ικανοτήτων που στηρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μας, για το Πανεπιστήμιο, είναι πώς μπορούμε αυτές τις πληροφορίες να τις διαθέτουμε όταν προκύπτει μια ερώτηση που πρέπει να απαντηθεί γρήγορα. Έχουμε ε, τα δεδομένα και τώρα εγώ προσπαθώ, ε, δουλεύω πάνω σε αυτό, να τα διαθέτω γρήγορα. Ε, αυτά βέβαια γίνονται όλα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν γίνει, ακόμα πάρα, έχουν γίνει πάρα πολλά, αλλά δεν υπάρχει συγκεκριμένη έκθεση που να δείχνει τι θα γίνει στην επόμενη φάση το πώς δηλαδή θα διαθέτουμε τις ε, πληροφορίες σε όσους ενδιαφέρονται. Ερωτήσεις τώρα παρακαλώ. Ευχαριστώ. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι ευρωπαϊκές ε, πρωτεύουσες, αυτή η πρωτοβουλία είναι πολύ σημαντική για πάρα πολλούς λόγους. Ε, με ενδιαφέρει κάτι. η ευκαιρία να ανανεωθούν οι πόλεις. Αναφέρεται στην ιστοσελίδα και δεν ξέρω αν μπορείτε να τοποθετηθείτε επ' αυτού. Κατοβίτσα, παραδείγματο χάρη, στην Πολωνία. Ε, θα ήθελε στο μέλλον να γίνει η πολιτιστική πρωτεύουσα και ανανεώνεται. Τι έχετε να πείτε επ' αυτού Άλλες ερωτήσεις, ο κύριος Χάιντερ Ένας από τους ε, πρώτους ομιλητές ε, ανέφερε ότι όταν πλέον λαμβάνεται μία απόφαση, δεν υπάρχει πλέον ε, πολιτική παρέμβαση και είναι όλοι ευχαριστημένοι. στη φάση που έχουμε την κριτική επιτροπή, εκεί υπάρχουν παρεμβάσεις πολιτικών. Προσπαθούν οι πολιτικοί να παρέμβουν. κυβερνήσεις ε, έρχονται και σας βρίσκουν, ε, σας λένε τις απόψεις τους ε, για να τις ακολουθήσετε. Αυτή είναι μια ερώτηση. Και μετά, σχετικά με τις έξι φάσεις εξελίξεων που πρέπει να επιτευχθούν, υπάρχουν κριτήρια που έχετε εντάξει στον κατάλογο ή είσαστε ικανοποιημένοι με όλα τα κριτήρια που ήδη υπάρχουν. Και επίση σε μία από τις ομιλίες άκουσα ότι έχουν γίνει σημαντικέ αλλαγέ στον προπολογισμό, προκύπτουν αλλαγέ στον προπολογισμό από την ώρα που προκυρήσεται ο διαγωνισμό μέχρι να οργανωθεί τελικά η πολιτιστική πρωτεύουσα. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, τότε τι ακριβώ κάνετε, η κυρία Βόρτ. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον που σας άκουσα, Μπεατρίς, από τη Λίβερπουλ, από την περιοχή μου. Πράγματι, η πολιτιστική πρωτεύουσα άλλαξε αυτήν την πόλη και υπάρχει. Αυτό είναι ορατό. Κάθε φορά που παίρνει κανείς ε, το τρένο ε, στο κεντρικό σταθμό στο Λίβερπουλ και πάρει μετά ταξί, όλοι οι ταξιτζίδες είναι πάρα πολύ φυλακοί. Ε, είναι εκπαιδευμένοι και είναι, λένε ότι είναι υπερήφανοι για την πόλη τους. Το έχω διαπιστώσει αυτό επανειλημμένα. Είχα πολλές συζητήσεις με τους οδηγούς ταξί στο Λίβερπουλ και αυτό προέκυψε ακριβώς λόγω της πολιτιστικής πρωτεύουσας. Ε, υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλές ε, συμπεριφορές που γίνονται ορατές της πόλεις. Δεν ξέρω τώρα αυτό που θα πω είναι ερώτηση, αλλά θα ήθελα κατά κάποιον τρόπο να πω ότι υποστηρίζω αυτά τα οποία κάνετε. Α, κάτι άλλο. Ε, σχετικά με την, το άνοιγμα, είπατε ότι πρέπει να ανοίξει η μελέτη δεν πρόκειται πια μόνο για ευρωπαϊκές πολιτιστικές πρωτεύουσες, πρόκειται για πολιτιστικές πόλεις και μεγάλες εκδηλώσεις, πώς ε, όλα αυτά μπορούν να επιφέρουν την αναγέννηση, να βοηθήσουν ώστε να αλλάξει ριζικά μια πόλη. Τώρα στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε ε, πόλεις πολιτισμού που εμπνεύστηκαν από πολιτιστικές ε, πρωτεύουσες Βλέπει λοιπόν κανείς μια φτωχή πόλη που πια τρέχει το δικό της το πρόγραμμα και ε, εκεί οι άνθρωποι νιώθουν ότι αλλάζουν, νιώθουν το δυναμισμό. Ο λόγος που δεν πήγα στη Ματέρα ήταν ε, γιατί μιλούσα σε ένα φόρουμ ανοιχτής οικονομίας στο Τορόντο, στον Καναδά. Αποφάσισα να πάω εκεί ε, και να γίνω η φωνή του πολιτισμού. Φωνή του πολιτισμού ως κινητήρια δύναμη της οικονομίας. Νομίζω ότι θα πρέπει ε, όλοι μας να είμαστε ε, πολύ περήφανοι για το τι κάνουμε εδώ, γιατί υπάρχει, μετακυλίεται αυτός, ε, αυτή η πρωτοβουλία, διαχέεται πολύ πιο μακριά Εγώ έχω μάθει πάρα πολλά για τις ε, πολιτιστικές ε, πρωτεύουσες. Τα έμαθα στο Open Economy Forum αλλά και σε άλλα βήματα όπου μου δίνεται ευκαιρία να μιλήσω και προσπαθώ να πω το πόσο καλά τα καταφέραμε ως ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα έλεγα να κλείσει ο κατάλογος των ομιλητών, να μπορούν να απαντήσουν ε, όλοι πριν φτάσει έξι ώρα. Συγγνώμη που ξαναζητάω το λόγο, αλλά επειδή δεν έχουμε πολλούς βουλευτές, γι' αυτό το κάνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μία ερώτηση προς τον δόκτωρα Γκαρσία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ χρήσιμη εισήγησή σας. Νομίζω ότι ε, δώσατε πολύ καλές ε, κατευθυντήρες γραμμές για τις ε, μελλοντικές πόλεις που ενδεχομένως να θελήσουν να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία της πολιτιστικής πρωτεύουσας. Μου, άρεσε, μου άρεσαν πάρα πολύ οι δείκτες που αναφέρατε. Η δική μου ερώτηση είναι, μήπως έχετε σκεφτεί σε αυτούς τους δείκτες να προσθέσετε και ένα δείκτη που να έχει σχέση με τις ε, περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Γιατί αυτό είναι ένα θέμα που καθίσατε όλο και πιο επίκαιρο ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Κοινοβούλιο. Έχουμε το Πράσινο Σύμφωνο ως ε, προτεραιότητα. Μήπως έχετε κάποια ιδέα τι θα μπορούσε να είναι αυτό τελικά. Yeah, who wants to start? Uh, uh, σε σχέση με τις ε, διαφορετικές ερωτήσεις ε, που υπευλήθησαν. Κοιτάξτε, ε, σχετικά με την τελευταία ερώτηση, θα ήθελα να σας πω το εξής. Το, θα άλλαζα κάτι στα κριτήρια και απαντώ ναι. Στα κριτήρια θα μπορούσα να αλλάξω κάτι και μετά θα... Mental dimension. Ε, ε, δηλαδή οι, διαδικασίες προσφοροδότησης να είναι ε, πιο σύντομες. είδαμε και στην αμερικάνικη περίπτωση την αντίστοιχη ότι μπορεί να γίνει αυτό. Επίσης όσον αφορά τα περιβαλλοντικά κριτήρια συμφωνώ και υπερθεματίζω. Δεύτερον, η global dimension είναι αυτή που μας ενδιαφέρει περισσότερο ε, σε αυτές τις διαγωνιστικές διαδικασίες, τις προσφορές. Ε, νομίζω ότι και αυτό είναι πολύ σημαντικό έτσι ώστε να τροφοδοτηθούν συζητήσεις και ε, διάλογος. Οι πολιτιστικές πρωτεύουσες είναι το καλύτερο φόρουμ για τέτοιου είδους συζητήσεις και για τοπική προοπτική ανάπτυξη και ε, γενικότερα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για το μέλλον. Ε, ε, η συνάδελφός μου τώρα να μιλήσει. Θα απαντήσω την ερώτηση ε, για την PSC και κατά πόσο υφιστάμεθα πιέσει, ε, Είναι πάρα πολύ δύσκολο να μας πιέσει κανείς γιατί είμαστε ανεξάρτητοι και ο στόχος μας είναι ένας και μόνο. Ο, ο κάλλιστος δυνατός θεσμός και η κάλλιστη δυνατή η υλοποίηση του θεσμού της πολιτιστική πρωτεύουσα. Βέβαια μετά ναι, είναι αλήθεια ότι μας στέλνουν ε, ε, mail ε, από ομάδες ας πούμε που θέλουν να επηρεάσουν λίγο τις αποφάσεις της ομάδας μας και αυτά από οργανώσεις πολιτών κλπ. Ε, στη διάρκεια της υλοποίηση, ναι, υπάρχουν πολλές προκλήσεις. και οι εθνικές κυβερνήσεις ε, βεβαίως έχουν υποστεί πίεση από μας και έχουν μάθει ότι εμείς είμαστε πάντα ε, με την πλευρά της ε, ομάδας που έχει κάνει την σωστή διαδικασία ε, του διαγωνισμού. Αυτούς θέλουμε να υποστηρίξουμε. Ευχαριστώ λέει η κυρία Μπέτρης Γκαρθία. Νομίζω ότι αυτά που ακούστηκαν ε, ήταν πάρα πολύ σημαντικά. Άλλη ερώτηση σχετικά με τους δείκτες και το φάσμα των δικτών. Κοιτάξτε, το ένα πλαίσιο δεν μπορεί να είναι ε, στεγανό. Πρέπει οπωσδήποτε να έχει την δυνατότητα κινητικότητας. Ε, γι' αυτό λοιπόν έρχομαστε σε επαφή με πανεπιστήμια, με ερευνητέ, όλοι συνεργαζόμαστε μεταξύ μα ε, έτσι ώστε να δούμε κάθε φορά ε, ποιο είναι ο τύπο τη πόλη, τη περιφέρεια και δεν μπορεί να υπάρχει μία λύση για όλα. Ναι, ενδεχομένως μπορούν να υπάρχουν κάποιοι κεντρικοί πυρηνικοί δείκτες και υπάρχουν και θέματα τα οποία είναι σημαντικά αλλά όχι πολύ σαφώς καθορισμένα όπως είναι ε, η ε, ευζοία ή όπως είναι ε, οι πολίτες πώς αντιλαμβάνονται αυτήν την ευημερία. Έχουν γίνει και αλλαγές. και εάν συγκρίνει κανείς ε, ε, τις πολιτιστικές πρωτεύουσες με πολύ μεγάλης, ε, μεγάλων διαστάσεων γεγονότα όπως ας πούμε είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε στα πλαίσια των πολιτιστικών πρωτεύουσών αυτά που έχουν γίνει στα πλαίσια του αθλητισμού γιατί για, του, τα Ολυμπιακά χωριά, για τους Ολυμπιακούς αγώνες αλλάζουν ακόμα και οι νόμοι, τα νομικά πλαίσια. Αυτό δεν μπορεί να γίνει για την πολιτιστική πρωτεύουσα. Ωστόσο, ναι, μπορεί να υπάρξει κάποια πίεση, αλλά και ε, είναι γεγονός ότι μπορούμε να εμπνευστούμε από κάποια άλλα από κάποιες άλλες εκδηλώσεις. Πλέον, μετά από τόσα χρόνια, ξέρουμε ότι η πρωτοβουλία είναι σωστή πρέπει να αναγνωρίσουμε τις επιτυχίες, αλλά θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνουμε και πιο εξεζητημένοι όσον αφορά την περιπλοκότητα και την αντιμετώπιση της περιπλοκότητας, ε, γιατί ε, εάν αρχίσουμε να θέτουμε ερωτήματα και να δίνουμε απαντήσεις ε, με, άσπρο, με όρους άσπρου μαύρου, τότε δεν διατρέχουμε τον κίνδυνο να αναπτύξουμε υπερβολικά πολλές προσδοκίες οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν. Και επίσης, επειδή όλες οι πόλεις δεν είναι ίδιες, μπορεί να δημιουργηθεί ε, η αίσθηση κακής κριτικής ε, απέναντι σε μια πόλη, η οποία υποτίθεται ότι δεν τα έχει καταφέρει τόσο καλά όσο μια άλλη πόλη. Ε, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε λοιπόν αυτή την έννοια της αποτυχίας, που δεν είναι αποτυχία, ε, και οπωσδήποτε ε, θα πρέπει να προωθήσουμε δείκτες που δεν θα ε, βασίζονται μονάχα στους, στα στατιστικά στοιχεία. Δεν υπάρχει μόνο άσπρο και μαύρο. Πολύ καλά τα είπατε και σχετικά με τον οδηγό του ταξί ε, νομίζω ότι αυτό πρέπει να είναι ένα σημαντικό στοιχείο για το μέλλον. Ε, και όσον αφορά την ε, περιφερειακή ικανότητα και το δυναμικό των πολιτιστικών πρωτευουσών, υπάρχει τέτοιο δυναμικό. Πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει καταρχήν και ένα όραμα για την ανάπτυξη της περιοχής. και αυτό σχετίζεται βέβαια και με την μοναδικότητα της, ε, του πολιτισμού στα πλαίσια της ε, πολιτιστικής ε, πρωτεύουσας και βεβαίως οι πολιτιστικέ πρωτεύουσε είναι πλέον πολλές ε, και ο διαγωνισμό δεν γίνεται μονάχα μεταξύ ε, ε, πόλεων της ίδιας χώρας αλλά και τελείως διαφορετικές χώρες γιατί ξέρουμε ότι πλέον θα είναι ταυτόχρονες οι πολιτιστικέ πρωτεύουσες σε διαφορετικές χώρες. Και ο θεσμός της πολιτιστικής πρωτεύουσας θα πρέπει να δώσει και κάποια όθηση στις πόλεις. Ε, και αυτή η όθηση βέβαια θα πρέπει, είναι δυνατή, αλλά θα πρέπει να γίνει με συνεκτικό τρόπο. Τέλος. Ευθύς εξ αρχής θα πρέπει το θέμα της πορείας της πόλης να το δούμε συνολικά και θέλω να επανέλθουμε σε ένα στοιχείο, σε μία από τις διαφάνειες υπήρχε το θέμα της βιωσιμότητας σε διάφορες διαστάσεις. Και νομίζω ότι ακριβώς αυτό είναι πολύ σημαντικό όταν συζητάμε για την κληρονομιά που μας αφήνουν αυτές οι δραστηριότητες. Ποιες είναι δηλαδή οι τάσεις οι οποίες παραμένουν στην πόλη και πώς μπορούν αυτές να χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια. και έτσι μπορούμε να έχουμε μια ευρύτερη συζήτηση που να τα συνδέει όλα αυτά με τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας. Ναι, και εγώ θέλω να πω ότι έχουν αλλάξει οι ρόλοι. Αν μαθαίνετε από τις προηγούμενες πολιτιστικές πρωτεύουσες, φροντίστε να μαθαίνετε από αυτές που είναι τώρα στην πορεία και όχι από τις παλιές. Αλλά έτσι καλώς μπορείτε να μάθετε από τα πάντα η ιστορία βοηθάει. Άμα δείτε την ιστορία, την κοιτάτε με τους σωστούς φακούς, θα μάθετε πολλά πράγματα. Πάρα πολύ ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι ήταν πολύ επικοδομητική αυτή η ακρόαση. Αποκομίσαμε πάρα πολλές ε, εντυπώσεις, επιβεβαιωθήκαμε σε πάρα πολλά. Ε, ε, εξετάσαμε το τι ακριβώς έγινε τα τελευταία χρόνια. Το κάνουμε αυτό συστηματικά ε, για να μπορούμε να έχουμε και τη σχετική εμπειρία. Ε, κατά τα άλλα όμως ε, θεωρώ ότι όλα αυτά είναι πάρα πολύ καλά. Αυτό που ενδιαφέρει είναι να ακούσουμε το τι ακριβώς έγινε καλά στο παρελθόν, που ακριβώς πρέπει να υπάρξει κάποια βελτίωση και ελπίζω από αυτά που αποκομίσαμε σήμερα ε, θα μπορούμε να ε, βγάλουμε αποφάσεις ε, για το μέλλον. Και θέλω να πιστεύω ότι η πολιτιστική πρωτεύουσα θα παραμείνει ένας φρέσκος θεσμός, θα χαρακτηρίζεται από βιωσιμότητα, Πολλοί να ανταλλάσσουν εμπειρίες, αν κάτι δεν πάει καλά, να γίνεται γνωστό, για να μην τα κάνουν και άλλοι τα ίδια τα λάθη. Νομίζω λοιπόν ότι έχουμε μια πολύ καλή πρωτοβουλία την οποία πρέπει να στηρίξουμε περαιτέρω και αυτό που ενδιαφέρει είναι οι πολίτες ε, στις διάφορες πόλεις να ενδιαφέρονται για τον ε, πολιτισμό ε, και να υπάρξουν και κάποιες αλλαγές, κυρίως όσον αφορά τα πολιτιστικά μακροπρόθεσμα, να δούμε τι μπορούμε να πετύχουμε και νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο ε, για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε αυτό το πρόγραμμα ε, να μπορέσουμε να επιτύχουμε πολλά σε διάφορες πόλεις. Ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα που μας είπατε και το πρώτο και το δεύτερο πάνελ και σας εύχομαι καλό βράδυ. Τα μέλη της Επιτροπής Πολιτισμού θα πρέπει να περιμένουν λίγο. Την επόμενη συνεδρίασή μας θα την έχουμε στις 20 Ιανουαρίου, Δευτέρα και Τρίτη 21 εδώ στις Βρυξέλλες και θα ήθελα... Τζούλη, παρακαλώ. Εκτός μικροφώνου, Τζούλη. Ε, θέλω να τελειώσω. Πες το τώρα, να τελειώνουμε. Ο λόγος που καθυστέρησα είναι γιατί είχα μία πολύ επίγουσα συνάντηση με κάποιους δικηγόρους. Έναν, ου, έναν επιμελητή εκθέσεων μουσείου από την Περσία. Κυρία είναι, είναι Ιρανή, καταδικάστηκε σε 10 χρόνια. Δούλευε για το Βρετανικό Συμβούλιο, για το British Council, για καθαρά διαπολιτισμικά προγράμματα. Είχα λοιπόν μία πολύ επίγουσα συνάντηση και θα ήθελα να ζητήσω από αυτή την Επιτροπή να οργανώσει μία ακρόαση για το θέμα αυτό. Ξέρω ότι έχουμε συμφωνήσει για πάρα πολλά, αλλά αυτό είναι επίγον και έκτακτη ανάγκη. Πρόκειται για καλλιτεχνικό παραγωγό ε, που ε, κανονικά ε, ασχολείται μόνο με τη δουλειά της, με εκθέσεις, καμία σχέση με πολιτική και τελικά καταδικάστηκε σε 10 χρόνια φυλάκιση. Ίσως μπορείτε να το συζητήσετε κάπως και να το βάλετε στη μέση διάταξη. Θα το εκτιμούσα πάρα πολύ αν το κάνατε αυτό. Ε, ίσως αυτό είναι μια περίπτωση για τα κατεπήγοντα στην Ολομέλεια. Νομίζω όμω και ότι ω ε, Επιτροπή Πολιτισμού κάτι πρέπει να κάνουμε. Η επόμενη συνάντησή μα θα είναι τον Ιανουάριο. Εντάξει, κάνει ένα πρόβλημα τον Ιανουάριο. Ίσως να το βάλετε ε, στα κατεπήγοντα της Ολομέλειας ε, του Δεκεμβρίου. Αν δεν τα καταφέρετε εκεί, τότε εντάξει πράγματι θα το συζητήσουμε με τους συντονιστέ στην επόμενη συνεδρία των συντονιστών ε, αν μπορούμε να το βάλουμε το θέμα στη μερική διάταξη. Ακρόαση λιγάκι δύσκολο, αλλά μπορούμε να γράψουμε μία επιστολή για να πιέσουμε. Και αυτό να το περάσετε και στα πρακτικά της σημερινής συνεδρίας ότι το έφηξα το θέμα. Στα διάφορα βάλτε το. Βέβαια είναι πολύ σημαντικό για να το αναφέρουμε στα διάφορα. Καλύτερα να το αναφέρουμε στην επόμενη συνεδρία των συντονιστών. Τελειώνοντας σήμερα, ε, θα ήθελα να σας ευχηθώ καλά Χριστούγεννα, γιατί είναι η τελευταία μας συνεδρίαση πριν τις ε, διακοπές των Χριστουγέννων και ελπίζω να σας δω υγιείς ε, και όλους ολομπρίο και δυναμικούς στην την επόμενη χρονιά. Να ξεκινήσουμε τον Ιανουάριο φρέσκοι και ζωντανοί. Σας ευχαριστώ πολύ.